Colleagues, let's get started. Uh, almost uh, minutes past the hour. Ε, είναι 9 και τέταρτο, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε. Πριν να μπούμε στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σας ανακοινώσω πως έχουμε μεταξύ μας μια αντιπροσωπεία για, της Κοινοβουλευτικής Εποπτικής Αρχής του Νοτιοαφρικανικού Κοινοβουλίου και παρακολουθούν τη σημερινή μας συνεδρίαση. Τους καλωσορίζω όλους ε, πολύ θερμά. Βρίσκονται εδώ αυτή την εβδομάδα μαζί με την γραμματεία τους υπό, μετά από πρόσκληση του Κοινοβουλίου μα, θα συναντήσουν τον Πρόεδρο Σούλτση καθώ και διάφορε επιτροπέ και αντιπροσωπείες. Είμαστε και πάλι μαζί κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού. Μία αντιπροσωπεία μα θα έχει επαφή μαζί με την, με την αντιπροσωπεία αυτή. Σα εύχομαι λοιπόν ε, κάθε επιτυχία στην ε, επίσκεψή σας στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Ε, μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα μας είναι το υπαριθμό 26. Πρόκειται για τον προϋπολογισμό του 2013, την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ο εισηγητής μας είναι ο Πίτερ Στάσνη από το ΕΛΚΑ. Πρόκειται για γνωμοδότηση για την υπεύθυνη Κοινοβουλευτική Επιτροπή που είναι βεβαίως η Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Πίτερ Στάσνη, έχεις το λόγο για να μας παρουσιάσεις τις ιδέες σου. Πρόκειται για το σχέδιο έκθεσης το οποίο έχετε στους φακέλους σας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τις ε, δημοσιονομικές διαδικασίες πριν να σας υποβάλω την εκθεσή μου. Καταρχήν, καθώς ήμουν εισηγητής ε, για τη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό πέρυσι και παλιότερα, ε, εκτιμώ το ρόλο της ε, Επιτροπής μας όσον αφορά την προώθηση και γνωτόμων ιδεών στον προπολογισμό. Το είδαμε πριν από λίγα χρόνια με την πρόταση για τα κέντρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τη θέσπιση μιας πλατφόρμας συντονισμού για τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, πράγμα που έχει να δεκτό στον τελικό προπολογισμό για το 2012. Βασιζόμενοι σε αυτά τα επιτεύγματα, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες πολύ νωρίς, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση και την εντολή για τον τριμερή διάλογο, ώστε να σηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητές μας και τις συστάσεις μας για τον προπολογισμό του επόμενου έτους στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. όντω. πρόκειται για την έναρξη μιας νέας δημοσιονομικής διαδικασίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτες η Κομισιόν συνέταξε την, το σχέδιο προπολογισμού για το 2014, πράγμα που θα εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες, ε, ε, εξηγώντα ε, συνεπώς και παρουσιάζοντας τις μεσονομικές μας προτάσεις σε αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά και στην εντολή για τον τριμερή διάλογο, καθώς και στη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό που θα γίνει το καλοκαίρι αυξάνουμε τις πιθανότητες να εισακουστούμε. Έτσι δεν είμαι μόνο εδώ για να παρουσιάσω αυτό το σχέδιο χνομοδότησης, αλλά ε, και για να ακούσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας προτεραιότητες και επιθυμίες για τον επόμενο χρόνο. Τη 9 Μαΐου πρώτη συνάντηση θα γίνει των εισηγητών ε, για τον προϋπολογισμό με την πρωτοβουλία του Γενικού Εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2013, τον κύριο Λαβία. Προσβλέπω στις, να ακούσω τις δικές σας απόψεις σήμερα. έτσι ώστε να έχω την εντολή, να, να σχηματιστεί εντολή για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας και στην Επιτροπή, στη σύσκεψη μάλλον, των δικών μας, ε, των εισηγητών περί προϋπολογισμού. Φυσικά θα λάβω υπόψη τις απόψεις αυτής της Επιτροπής τονίζω τις σχέσεις ε, τις εμπορικές με τις γειτονικέ χώρες, τη διατήρηση των, ε, των ε, κονδυλίων για τα μέσα εταιρική συνεργασία, καθώς και για τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις που είναι σημαντικές για τις σχέσεις της Ένωσης. Επίσης, χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Πολιτικής για το 2013. Ε, και τώρα θα ήθελα να ακούσω απόψεις των σκιωδών και των μελών της Επιτροπής μας, ε, τα σχόλιά σας για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης ή σε σχέση με τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, Μπέρτε Λάγκε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε... Ε, κύριε Σιγητά, σας ευχαριστώ για την υποβολή της νομοδότησής μας. Ζητήσατε να υποβάλουμε νέες ιδέες, το κάνατε αυτό με εξαιρετικό τρόπο και πολύ σωστά. Εγώ θέλω ένα πράγμα μόνο να προσθέσω. Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να διατηρήσουμε τα όσα έχει ήδη επιτύχει η Επιτροπή μας, που έχει ήδη παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού εχθές το απόγευμα και μιλά για μια αύξηση 6,8% του όγκου του προϋπολογισμού. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξαν ε, πολλές δεσμεύσεις στην ε, διαρθρωτική πολιτική και που τώρα πρέπει να τηρηθούν. Πρέπει να γίνουν δηλαδή πληρωμές. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να αποφύγουμε, γιατί δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι του προπολογισμού θα είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Εφόσον λοιπόν έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, θα πρέπει και να τις σεβαστούμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιμείνουμε για περαιτέρω ε, προγράμματα, αλλά καλύτερα είναι να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά που έχουμε ήδη εγκρίνει όσον αφορά το πολιτικό μας πρόγραμμα και την πλατφόρμα για τα μικρομεσαία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε για την κοινοτική πολιτική να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ακόμη καλύτερα όσον αφορά τις επιτυχίες των, ε, του πιλωτικού προγράμματος. Υπάρχουν ήδη δομές ε, που λειτουργούν και που αφορούν ένα ισότιμο δίκαιο εμπόριο. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το τονίσουμε. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του εισηγητή. Thank Κάποιος από την Επιτροπή για αυτό το σημείο. Όχι. Ναι, ναι. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ να μας πείτε το όνομά σας, παρακαλώ, για τα πρακτικά. Καλημέρα σας. Λέγομαι Ιφαν Μποκοβίτιτς από την DG Trade, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Νομίζω πως ο εισηγητής... Yeah. The difficult issues we will have in τόνισε τις δυσκολίες που θα έχουμε στην ε, χρήση τη δημοσιονομική του 2013 γιατί η Επιτροπή ενέκρινε εχθές την ε, ε, χρήση του 2013 και είπαμε ότι είναι δύσκολο, υπόθηκε και χτες, τόσο γιατί είμαστε σε δύσκολο οικονομικό πλαίσιο, αλλά και επειδή ε, ο προπολογισμό του 2013 είναι ο τελευταίος χρόνος της, ε, του πολιατού δημοσιονομικού σχεδιασμού που πράγμα που επιβάλλει τη τήρηση των δεσμεύσεων, την κάλυψη των δεσμεύσεων που είχαν αναλυφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Καθώς θα διαβάζετε το σχέδιο προπολογισμού θα διαπιστώσετε ότι Έχουμε λάβει υπόψη την ε, λιτότητα υπό την οποία ζούμε όλοι, όμως έχουμε εντοπίσει τομείς προτεραιότητες που ορίζονται και ορίζονται και στη στρατηγική ανάπτυξη για το 2020 και ως προς αυτό θα ήθελα να τονίσω πως 62,5 δις ευρώ αφιερώνονται στην ανάπτυξη, στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Final remark. Τελικές ε, καταληκτήρες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ στον συνάδελφο και την Επιτροπή για τις παρατηρήσεις τους. Και άκουσα χτες και τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι. Ε, και βέβαια υπάρχουν ε, αντιφάσεις, αλλά νομίζω ότι αυξάνουμε κάτω από την πληθωρισμό, άρα κατά βάση μειώνουμε τον προπολογισμό μας. Και με ευχαρίστηση είδε ότι οι αυξήσεις βασικά αφορούσαν την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα, το, την παιδεία, ενώ εδώ έχουμε καινοτομία. Εδώ έχουμε διψήφια νούμερα και εδώ συμφωνούμε γιατί αυτές είναι οι επενδύσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη και τη μελλοντική απασχόληση. Καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι εύκολο και η Κομισιόν είπε ότι πρόκειται για να μείνει προπολογισμό, αλλά ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τις, τις συνειλημμένες υποχρεώσεις μας. Πάντως, να σας πω με ευχαρίστησή μου ότι κινούμεθα, κινούμεθα σταδιακά. Ήδη υπάρχουν κάποια προγράμματα που είναι θεσπισμένα και λειτουργούν, ή δεν τα ανέφερα, υπάρχει και ένα με τη Μεσόγεια όπου οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν ως μέντορες για τις ε, βορειοαφρικανικές επιχειρήσεις για τις ε, περιοχές γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω πως όπως και στο παρελθόν αυτό το σχέδιο κοινή λογικής θα βρει γόνιμο έδαφο και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και θα προχωρήσει προς όφελες των πολιτών και των δύο όχθεων της Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, calendar. Σας ευχαριστώ πολύ. Ημερομηνίες. Εδώ έχουμε ονομοδότηση που πάει σε άλλη επιτροπή, την Επιτροπή Προπολογισμού, οπότε το χρονοδιάγραμμά μας ε, είναι υποπίεση χρονική. Έχουμε λοιπόν προθεσμία για υποβολή τροπολογιών την επόμενη, την, στις 3 Μαΐου. 3 Μαΐου το απόγευμα, στις 6. Και στην επόμενη μας τακτική συνεδρίαση θα εξετάσουμε το σχέδιο με τις τροπολογίες. Πάμε στο σημείο 27. Κατάσταση όσον αφορά τις προσχωρήσεις στον ΠΟΕ. Εδώ έχουμε παρουσίαση της Κομισιόν και συζήτηση στη συνέχεια. Όπως ξέρετε, ο ΠΟΕ ε, γίνεται παγκόσμιος οργανισμός. Στην ουρά περιμένουν, σύμφωνα με τη σημειώσεις μας, το Καζακστάν, το Αζερβαϊτζάν, το Τατζικιστάν και το Λάος. Και επίσης, στην τελευταία υπουργική διάσκεψη που έγινε το Δεκέμβριο στη Γενέβη, αποφασίστηκε η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών του 2002 για την προσχώρηση των ε, λιγότερων αναπτυγμένων χωρών ε, στον ΠΟΕ. Οι συστάσεις αυτές όμως ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά θα πρέπει να παρουσιαστούν τον Ιούλιο, μέχρι τον Ιούλιο φέτος. Να ακούσουμε λοιπόν την Κομισιόν αν υπάρχουν πρόσφατες εξελίξεις και πώς αξιολογούν την κατάσταση. Ο Παύλο Γκαρσάτη θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να σας ενημερώσω για τις προσχωρήσεις των ΠΟΕ. Όπως είπατε, Διακόπτει ο πρόεδρος. Ησυχία. Τι γίνεται εκεί. Should be held Και καθίστε παρακαλώ. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει να βλέπω να στέκονται όρθιοι σε αυτή τη συνεδρίαση. Είναι θέμα σεβασμού για, προς τους ομιλητές ιδιαίτερα σε σχέση με τους φιλοξενούμενους από άλλα θεσμικά όργανα. Λοιπόν, Επιτροπή, συνεχίστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως έλεγα, λοιπόν, οι προσχωρήσεις, όπως και εσείς αναφέρατε, στον ΠΟΕ, είναι όλο και περισσότερο ένας παγκοσμιοποιημένος πλέον οργανισμός ε, για όσον αφορά την εντολή του. Καλά μαντάτα αυτά σε σχέση με την πολυμερή ε, εμπορική υποστήριξη στρέφονται στον ΠΟΕ διάφορα κράτη για την ρύθμιση θεμάτων παγκοσμίου εμπορίου όλο και περισσότερο. Όπως είπατε πρόοδος έγινε το 2011, σημαντική πρόοδος. Φυσικά όμως υπήρξε και ένα ορόσημο της Ρωσίας που εντάχθηκε στον ΠΟΕ Ουσιαστικά δηλαδή η νομική προσχώρηση της ε, Ρωσίας θα επιτευχθεί το αργότερο στις 21 Αυγούστου 2012. Η διαδικασία επικύρωσης ακόμα βρίσκεται υπό εξέλιξη στη Ρωσία. Και αυτό θα είναι ένα σημαντικότατο στοιχείο, ένα σημαντικός νέος εταίρος της οργάνωσής μας. Πέρα από αυτό είχαμε ένα σημαντικό ε, γείτονα εταίρο το Μαυροβούνιο μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και αναμονή και σε σχέση και με την Ουκρανία που ε, επετεύχθη η προσχώρηση της στον ΠΟΕ τελευταία, στην τελευταία φάση και το με το, την επικύρωση του πρωτοκόλου θα εγγραφεί και αυτή η Σαμόα και εκείνη. Είναι ένα θέμα που λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και συμφέρον σε σχέση με την οργάνωσή μας. Και τέλος η Βανουάτου, όπου έχουμε μια αξιοπερίεργη διεργασία εδώ είχε ήδη εγκρίνει να προσχωρήσει το 2001, αλλά δεν επικυρώθηκε η διαδικασία του πρωτοκόλου προσχώρησης. Επανήλθαν το 2008, ξανάρχισαν νέες διαπραγματεύσεις, νέο πρωτόκολλο, νέα έγκριση πρωτοκόλου 2000 από πλευράς ΠΟΕ, μια καθυστέρηση σε σχέση με την προθεσμία από πλευράς Βανουάτου για την επικύρωση αυτού του πρωτοκόλου λόγω εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων και τριβών θα δούμε πώς αυτή η μικρή νησιωτική χώρα θα προχωρήσει. Σε σχέση με προοπτικές για το 2012 τώρα, οι τέσσερις προτεραιότητες που ταυτοποιήθηκαν, που εντοπίστηκαν επίσημα από τα μέλη, από με τη γραμματεία του ΠΟΕ, και φυσικά αυτό δεν παρακολεί το να προχωρήσουν άλλα θέματα προσχωρήσεων. Είναι το θέμα του Καζαχστάν, της Σερβίας, Λάος και η Εμένης. Ε, και σε σχέση με αυτές τις ε, επιμέρους προσχωρήσεις, η διαδικασία για την προσχώρηση είναι συγκρίσιμη. Θα ε, διαιρούσα, θα κατένιμα σε τρεις ομάδες τις ε, χώρες αυτές. Δυτικά Βαλκάνια πρώτον, λόγω και της σημασίας που έχει αυτή η περιφέρεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε όπως είπα τη Σερβία που έχει εγγραφεί στον κατάλογο των χωρών προς υποπροσχώρηση που θα πρέπει να επιτευχθεί αν είναι εφικτό μέχρι, το 2000, μέχρι και το τέλος του 2012. Η Σερβία έχει προχωρήσει αρκετά στις διμερείς ε, διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των αγορών. Όμως δυστυχώς έχουν θέμα που εκρεμεί και πάλι εδώ με την, για την Κράινα όπως ε, και σε σχέση με διάφορα θέματα διαπραγμάτευσης ε, είναι δύσκολη αυτή η πτυχή και υπάρχουν προβλήματα. Πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό με την διαπραγμάτευση FDA η ίδια διαδικασία όπως για το Μαυροβούνιο, τα θέματα δηλαδή, δύσκολα θέματα για την πρόσβαση στην αγορά μέσω FDA να μπορούσαν να ρυθμιστούν και διμερούς πρωτοκόλου με, το, με τον ΠΟΕ. Η προσχώρηση της Σερβίας τώρα στο πολυμερές πλαίσιο, το μόνο νομικό πρόβλημα που έχουν είναι το πρόβλημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Τι γίνεται εδώ θα πρέπει να αναθεωρήσουν το νομικό τους πλαίσιο για να προσαρμοστούν σε σχέση με το εσωτερικό νομικό ε, πλαίσιο της Σερβίας είναι το μόνο εμπόδιο που εκκρεμεί ακόμα. Βοσνία Ζεγοβίνη, άλλη σημαντική αυτή βαλκανική χώρα με προοπτική ένταξη. Αυτή δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο η Σερβία. Αυτό οφείλεται και στη διαφορετική πολιτική κατάσταση που ε, υπάρχει στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ελπίζουμε ότι η τεχνική πρόοδος θα επιτευχθεί το 2012 ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η προσχώρηση του, από του χρόνου 2013. Η δεύτερη ομάδα είναι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, η δεύτερη ομάδα χωρών. Δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν δύο λιγότερο ανεπτυγμένες χάρες που αναμένουν να ενταχθούν το 2012. Η μία είναι το Λάος που έχει προχωρήσει πολύ και με θετική τεχνική υποστήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις είπα τους συνήθεις χορηγούς αλλά και με σημαντική εμπλοκή και προσπάθειες της Κίνας προωθώντας την ένταξη αυτής της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας. Αυτό δείχνει και το νέο ρόλο της Κίνας στον ΠΟΕ υπό αυτή την πτυχή. Εμείς και πάλι μπορούμε να πούμε ότι το Λάος αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες σε σχέση με την ολοκλήρωση διαδικασιών αλλά θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα και να ρυθμιστούν. Το ίδιο ισχύει για την Ιεμένη για την οικονομική ένταξή της στον ΠΟΕ για πριν από μερικά χρόνια που μπορούσε να προωθηθεί. Για κάποια χρόνια όμως δεν μπόρεσε να σημειωθεί πρόοδος. Τώρα που η πολιτική κατάσταση σταθεροποιήθηκε, τώρα που η πολιτική κατάσταση σταθεροποιήθηκε, συγγνώμη, μπορούν με πλήρη όθηση να προχωρήσουν, ζητεί μηδενικούς δασμούς ε, όσον αφορά χαλιβουργικά προϊόντα στην ε, η η Ουκρανία. Διαρωτάται κανείς ποιο μπορεί να είναι το εμπορικό συμφέρον να ζητεί κάτι Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά όμως ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία επί του θέματος υπήρξε αρκετός βαθμός ελαστικότητας, ευελιξίας έναντι της Ιεμένης υπάρχει προθυμία κάποιας μεταβατικής ε, περίοδου που θα εγκρινόταν, πράγμα το οποίο ε, δεν ε, τίθεται ως προοπτική για άλλες χώρες υπό προσχώρηση, υπό ένταξη. Τώρα, σε σχέση με την Υπουργική Διάσκεψη του προηγουμένου Δεκεμβρίου υπήρξε συμφωνία να υπάρξουν νέες κατευθυντήριες γραμμές που θα διαπραγματευτούμε και θα εγκριθούν σε σχέση με τις υφιστάμενες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως εμπλέκεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αφενός η θέση μας είναι να διασφαλίσουμε οπωσδήποτε ότι αυτές οι χώρες θα μπορούν να τύχουν μιας ε, χωρίς προβλήματα διαδικασίας ε, προσχώρησης, ε, με βοήθεια υποστήριξη που θα τους δοθεί, με μεταβατικές περιόδους, με ήπια πίεση που θα ασκηθεί για την για τα θέματα πρόσβαση στην αγορά. Συμφωνούμε να υπάρξουν βέλτιστες προδιαγραφές ε, για την πρόσβαση στις αγορές σε σχέση με συγκεκριμένα αγαθά. Ταυτόχρονα μεριμνούμε όμως οι προσχωρήσεις των χωρών, των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών να μην ακολουθούν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία στην προσχώρηση αυτών των χωρών, διότι η διαδικασία μεταρρύθμισης που είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο αγαθό σε σχέση με την προσχώρησή τους στον ΠΟΕ, η εσωτερική διαδικασία μεταρρυθμίσεων μπορεί να υπονομευθεί και έτσι θα μπορούσε να απολεστεί ένα από τα πιο σημαντικά ωφέλη διαπραγματεύσεις που διεξάγονται σε σχέση λοιπόν με αυτές τις χώρες, το πιο σημαντικό και πιο ενεργό κράτος προς ένταξη είναι το Καζαχστάν. Γιατί είναι σημαντικό το Καζαχστάν, διότι είναι, αποτελεί σημαντικό τμήμα της Τελωνιακής Ένωσης ε, σε σχέση με τη Ρωσία. Και ολοκληρώσαμε διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή για ε, το κόστος, το, τα, δασμολόγια για τις εισαγωγές. Υπάρχει συμφωνία σε σχέση και συμφωνεί με το, το Καζαχστάν διμερός όσον αφορά τον ΠΟΕ. Θα πρέπει αυτά τα θέματα να, να διαπραγματευτούμε σε σχέση με την Τελωνιακή Ένωση. Μετά την ολοκλήρωση των διμερών διαβουλεύσεων και την ένταξη του Καζαχστάν στην Τελωνιακή Ένωση με τη Ρωσία και την Μπελαρού στη Λευκορωσία θα πρέπει αυτά τα θέματα των δασμών να τύχουν διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ΠΟΕ. Θα πάρει χρόνο αυτό. Είναι ένα περίπλοκο ε, ζήτημα. Θα πρέπει να ζητηθεί αντιστάθμιση για κάποια ζητήματα όπου έχουν αυξηθεί οι δασμοί και τα τέλη με αρκετές μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ιστερότερα κατά τη διάρκεια του 2012 η διαδικασία προσχώρησης του Καζαχστάν να μετατεθεί για υστερότερα ακόμα. Ένα άλλο θέμα που εκκρεμεί είναι το θέμα των δασμών εξωτερ... για τις εξαγωγές. Έχουμε συμφέροντα στην περιοχή όπως και σε σχέση και με τη Ρωσία όσον αφορά τη στρατηγική μας για τις πρώτες ύλες διαπραγματευόμαστε σε σχέση με τις δεσμεύσεις για σημαντικά θέματα πρώτων υλών όσον αφορά και το Καζαχστάν. Σε σχέση με τις εσωτερικές επενδύσεις και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στο Καζαχστάν, το πρόβλημα που πρέπει εκ του σύνεγγυς να εξεταστεί περισσότερο είναι τα μέτρα σε σχέση με τις επενδύσεις και επενδυτές. Αντιγράφουν κάποιες ε, μη θετικές ε, πρακτικές από άλλες γειτονικές τους χώρες και πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό με ιδιαίτερη προσοχή. Υπήρξε κάποια πρόοδος ε, ή τουλάχιστον σε σχέση με την, ε, την Αλγερία εδώ δυστυχώς από ό,τι μπορούμε να πούμε η πολιτική αυτή κινητοποίηση όσον αφορά την ε, Αλγερία δεν επαληθεύεται σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στο τραπέζι. Παράδειγμα, η νέα προσφορά σε σχέση με του να υπάρξει ένα 49% συμμετοχής από αλλοδαπούς όσον αφορά επενδύσεις στην Αλγερία αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα καλωσορίζαμε και θα μπορούσαμε να καλοδεχθούμε στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την ένταξη αυτής της χώρας στον ΠΟΕ. Άλλα θέματα ένταξης που ε, κινητοποιούνται κάποιες χώρες είναι τα θέματα των Σεϊχελών και ε, το θέμα που αφορά τις Μπαχάμες. Εδώ τουλάχιστον για την δυνατότητα να δοθεί υποστήριξη σε σχέση με αυτές τις χώρες δεδομένης της ειδική μας σχέσης με αυτές λόγω της οικονομικής, των οικονομικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών εταιρική σχέσης που έχουμε με αυτές. Φυσικά θα μπορούσα να επεκταθώ περισσότερο, προτιμώ να υπαρκεστώ σε αυτά τα σχόλια και να παρέμβουν οι ευρωβουλευτές αν έχουν κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νόμιζα ότι μιλούσατε για το εμπόριο, όχι για τον τουρισμό, Τέλο πάντων. Νομίζω ότι ανάμεξα αυτά τα δύο. Λοιπόν, μπορεί τώρα να αρχίσει η συζήτηση. Παρακαλώ τους βουλευτές, όποιον θέλει το λόγο, κύριο Στάσνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας, να διευκρινίσω, γιατί δεν κατάλαβα καλά αν μιλούσε για την Αλγερία, για την Ιγυρία εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ε, μάλλον για την Ιγυρία μιλάει, αλλά νομίζω ότι άκουσα Αλγερία. Επίσης. Any other question? Bernd Για το ΠΟΕ. Ναι, σας ευχαριστώ. Η διαδικασία είναι αυτή που περισσότερες χώρες ε, θέλουν να ενταχθούν στον ΠΟΕ ή ε, βρίσκω ότι είναι καλό αυτό ως πρωτοβουλία. Διότι φυσικά το διεθνές πλαίσιο για το εμπόριο από πλευράς ΠΟΕ είναι το πιο βιώσιμο και αηφόρο πρότυπο. Καλό είναι ότι και συμμετέχουν η Ρωσία, η Κίνα και θα συμμετέχουν και πολλά άλλα κράτη, ακόμα και όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτηση προς την Επιτροπή. Πώς εκτιμάτε το δυναμικό δυναμικό που μέσω αυτής της ένταξης της Ρωσίας, της Κίνας αλλά και πολλών άλλων μικρότερων χωρών έχει επισημανθεί ότι με αυτές τις μικρότερες χώρες υπάρχουν ειδικέ σχέσεις σε σχέση με μεγαλύτερες χώρες. Μέσω αυτών των θεμάτων η δυναμική του ΠΟΕ θα μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο ή αυτός ο πρόσθετος αριθμός κρατών μελών θα είναι τροχοπέδι για τη διαδικασία μεταρρύθμισης και την διεύρυνση και συνέχιση των συζητήσεων για τον γύρο της Δόχα. Για την Ουκρανία έχω και εγώ ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Είπατε ότι η Ουκρανία προσελκύει και πάλι την προσοχή υποβάλλοντα ενστάσεις για την προσχώρηση του ΛΟΣ και της Ιεμένη. Αν σας κατενόησα, καλώ. Το ίδιο έκανα και πέρυσι με το Μαυροβούνιο. Δηλαδή τελικά τι είναι, θα δημιουργήσουν προβλήματα, πώς το βλέπετε, θα είναι ταραχοποιή του ΠΟΕ. Βλέπουμε ότι ο ΠΟΕ γίνεται μια όλο και πιο οικουμενική οργάνωση. Και οι κανόνες του επομένως. Θέλω την άποψη του εκπροσώπου της Κομισιόν ως προς το βαθμό στον οποίο ο αυξανόμενος αριθμός προσχωρήσεων θα μπορούσε να επηρεάσει την δυνατότητα και ικανότητα του που ένα ε, δίνει αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά την νομοθετική του αρμοδιότητα, αλλά και τον εποπτικό του ρόλο, την επίλυση των διαφορών αυτές τις εξελίξεις, πώς τις εκτιμάτε. Σε σχέση, επαναλαμβάνω, με τη δυνατότητα του ΠΟΕ να φέρει σε πέρα στα καθηκοντά Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές για τα ενδιαφέροντα ερωτήματά τους. Θα απαντήσω στη, με τη σειρά τα ερωτήματα όπως μετέθησαν. Αλγερία έλεγα, ε, γιατί η Νιγηρία είναι ήδη μέλη του ΠΟΕ. Ναι, συγγνώμη, μέλος του ΠΟΕ. Η Αλγερία έχει ακολουθήσει ένα περίεργο μονοπάτι. Ήταν μέλος του ΓΚΑΤ, μετά συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ε, του ΠΟΕ. Δεν προσυπέγραψαν όμως στο τέλος. Είναι δηλαδή σε εξέλιξη η διαδικασία, αλλά έτσι όπως βλέπουμε να εξελίσσεται η κατάσταση ιδίω της οικονομίας στην Αλγερία, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η προσχώρηση της χώρας στον ε, ΠΟΕ. Πρέπει να αποδείξει ακόμα ότι μπορεί να πληρώσει όλες τις προϋποθέσεις. Όταν η Ρωσία, η Σαμόα και το Μαυροβούνιο επηρεάσει, θα έχουμε, ε, συγγνώμη, υπογράψουν, θα έχουμε 156 χώρες πλέον. Ο πρόεδρος έκανε δύο ερωτήσεις, ε, μάλλον ο πρόεδρος και ένας ε, βουλευτής για το κατά πόσο αν υπάρχει ένα πρόβλημα ή αν είναι ευκαιρία το ότι αυξάνονται δηλαδή οι προσχωρήσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι ευκαιρία οι προσχωρήσει αυτές και όχι μόνο ευκαιρία, αλλά αυτό προσδίδει μεγαλύτερη νομιμοποίηση στον ΠΟΕ, που είναι μια οργάνωση όπου όλοι έχουν λόγο, σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς που μια χώρα με την ψήφο της μπορεί αν θέλει να σπάσει τη συνένεση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, σε ό,τι αφορά την πρόοδο επί της ατζέντα της Ντόχα, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση πάντα με τον αριθμό των μελών. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ατζέντα της Ντόχας μέχρι τώρα, αλλά αυτό δεν οφείλεται στα νέα μέλη που έχουν προσχωρήσει. Αλλά στις δύο μεγάλες οικονομικές δυνάμεις σήμερα στον κόσμο, την Κίνα και τη είπα δηλαδή. Τούτο λεχθέντος δεν υποτιμώ τη σημασία που έχει το ότι η Ρωσία αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως μέλος των χωρών BRICS και στο πλαίσιο του ΠΟΕ στα εμπορικά ζητήματα. πριν από καμιά δύο μέρε είχαμε την υπουργική διάσκεψη ε, των υπουργών εμπορίου ε, του G20 που με ένα, ε, μια μικρή τη δήλωση η Ρωσία συντάχθηκε πλήρως με τις, χώρες, τις άλλες χώρες BRIC. Τώρα αυτό πώς θα εξελιχθεί δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Η Ρωσία έχει προσχωρήσει τον ΠΟΕ ως αναπτυγμένη χώρα. Άρα μπαίνει σε διαφορετική θέση από τις τρεις εναπομένες χώρες των χωρών BRIC, ή BIC δηλαδή, που είναι ανάπτυξη ακόμη χώρες. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις τώρα για τη διευκόλυνση του εμπορίου στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχα. Η Ρωσία εκεί φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πολύ για τη διαμετακόμιση και ιδίω ε, την οδική διαμετακόμιση, αλλά θέλει να εφαρμοστεί και στους αγωγούς η διαμετακόμιση ως ε, μια τελωνιακή οργάνωση που βασίζεται κυρίως στην ίσπραξη και όχι τόσο στη διευκόλυνση, η Ρωσία θα πρέπει να κάνει κάποιες προσαρμογές. Συνολικά όμως, Η Ρωσία πρέπει να τηρήσει όλους τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που διέπουν από την ένταξη Τον ΠΟ και αυτό είναι θετικό. Δεσμεύεται. Σε ό,τι αφορά τώρα την επίλυση διαφορών και το ρόλο του ΠΟΕ, είναι σαφές ότι η Ρωσία θα είναι ένας ενεργός χρήστης, όπως όλες οι χώρες βέβαια ε, του ΠΟΕ. Και για να συνοψίσω. The uh, cost benefit balance uh, uh, is αν ε, ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά, νομίζω ότι τα υπέρ υπερτερούν, ε, πλεονεκτούν. Έχουμε και κάποια ειδικά συστήματα, έχουμε και το, ε, το καθολικό σύστημα της διακυβέρνησης. Θα παρακολουθούμε τα πράγματα και βέβαια θα ερχόμαστε εδώ για να συζητάμε τα πράγματα και γενικότερα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις προσχωρήσεις νέων χωρών. Για την Ουκρανία τώρα. Ήδη δημιουργούσε προβλήματα. Άρχισε να τα δημιουργεί μόλις εντάχθηκε ε, με το Μαυροβούνιο, όπως είπατε. Και πέρυσι με τη Σαμόα δημιούργησε πρόβλημα, της νήσου Σαμόα υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική στάση της Ουκρανίας. Λέει πολλά πληρώσαμε για να γίνουμε μέλος του ΠΟΕ και τώρα ζητάμε και εμείς σε αντάλλαγμα πολλά από τους άλλους. Κάποιες φορές μας εκπλήσει το επίπεδο των δεσμεύσεων που ζητούν από μη ανεπτυγμένες χώρες. Υπάρχει πάντως μια διαδικασία στην Γενέβη αυτή τη στιγμή για να τεθούν πιέσεις όχι μόνο διμερώς αλλά και στο πλαίσιο του ΠΟΕΝ για την Ουκρανία να σκεφτούν λοιπόν πιέσει στην Ουκρανία στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που συνεδριάζει και ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Ιεμένη και ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Λάος με την Υποεπιτροπή αυτή και με τον διαπραγματευτή τον Ουκρανό για να δημοσιολαβήσουν ώστε να λυθεί το πρόβλημα ο ήχους που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής είναι ότι ίσως αυτές οι πιέσεις σε κάποιο βαθμό φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, διότι υπάρχουν συνεχείς διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις λιγότερα αναπτυγμένες χώρες που θεσπίσουν συγκεκριμένα benchmark, συγκεκριμένα ε, συγκριτικά όρια αναφοράς για τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Και όλα αυτά βέβαια έρχονται σε αντιπαράθεση με την στάση της ε, Ουκρανίας. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτά τα πρώτα χρόνια φαίνεται να σκέφτεται κάπως διαφορετικά η Ουκρανία. Ε, ε, Έχετε άλλες ερωτήσεις? Να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του εκπροσώπου της Επιτροπής εδώ. Όχι. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για αυτή την πολύ ενημερωτική... Uh, we have to make a small suspension of our meeting because next... Νομίζω ότι τώρα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Στις 10 όμως θα ψηφίσουμε. 10 ε, λεπτά διάλειμμα λοιπόν για να ξεκινήσουμε στις 10 της ψηφοφορίας.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 πιστεύει. space.

Θα ξεκινήσουμε ψηφίζοντας για μια διαδικαστική απόφαση. Που σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν εχθές στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών αφορά τον κανονισμό για εξαιρετικές προτιμήσεις για το Πακιστάν. Όπως ξέρετε, πέρσι υιοθετήσαμε τις ε, εκθέσεις ε, ίντα στην Ολομέλεια, αλλά δεν υπήρξε πρόοδο στον ΠΟΕ και έτσι αναστέλει η διαδικασία. Εν τω μεταξύ όμω υπήρξε πρόοδο ε, στον ΠΟΕ και η Κομισιόν ζήτησε από το Κοινοβούλιο να επαναλάβει τη διαδικασία εκεί όπου είχε σταματήσει πέρσι. Εχθέ οι συντονιστέ λοιπόν αποφάσισαν να επαναλάβουν τη διαδικασία και να ζητήσουν από την ολομέλη εντολή για να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Κομισιόν εν ώψη σύναψη μια συμφωνία πρώτη ανάγνωση για αυτό το φάκελο. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεκινήσει άτυπε διαδικασίε με τα άλλα θεσμικά όργανα, αναμένοντα ένα αναμονή μάλλον τη απόφαση τη Ολομέλεια. Ξεκινάμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Uh, να δούμε την απόφαση λοιπόν ε, που θα πρέπει να λάβουμε. Να ζητήσουμε από την Ολομέλεια να επαναλάβει τη διαδικασία για αυτό το θέμα στο σημείο που είχε σταματήσει πέρσι και να ζητήσουμε την έναρξη τριμερού διαλόγου με το Συμβούλιο ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία πρώτη ανάγνωση. Δεύτερον, να ξεκινήσουμε άτυπτο διάλογο με το Συμβούλιο και εν αναμονή της, ε, της ε, έγκρισης. Λοιπόν, έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζουμε, ψηφίζουμε. And the vote is... The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. The is closed.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 Να ζητήσω λοιπόν από τους, ε, από τους τη διάσκεψη των να τοποθετήσουν το ψήφισμα στην ε, επόμενη μερίσια διάταξη και τώρα... Θα πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ξέρετε ίσως ότι έχει επιτευχθεί συμβιβαστική στο Συμβούλιο μεταξύ των κρατών μελών, οπότε ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να βρεθεί και συμβαστική ανάμεσα σε εμά και το Συμβούλιο. Άλλη ερώτηση τώρα του για την Κομισιόν. Να, να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο. Λάγκε, Ντάβιντ, έχετε το κείμενο στους φακέλους σας. Πρέπει να ψηφίσουμε για αυτή την προφορική ερώτηση που έχουν υποβάλει αυτοί οι συνάδελφοι. Ε, <clears throat> ψηφίζουμε. And the vote is closed. It was adopted by 21 votes. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ και μία κατά. Συγχαρητήρια στους συντάκτες της προφορικής ερώτησης. The draft report on the regulation Περνάμε τώρα στο σχέδιο έκθεσης ε, για κανονισμό που θεσπίζει γενικές διατάξεις για την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς τρίτες χώρες. Ε... <coughs> Η μας είναι ο κύριος Καζάκ. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για την έκθεση Καζάκ. Ξεκινάμε με τις τροπολογίες. Τροπολογία ένα. Uh, the vote is open. Uh, no, please. It's an open vote. So who's in favor? Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. Ε, τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. 67. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 και 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Where is 72? Yeah. Ah, 72. Yes. 72. 72. Υπέρ, κατά. Εποχές εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία 73 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Πολ Μέρφυ. Not on the Δεν βρίσκεται στον κατάλογο των σοσιαλιστών. Ναι, αλλά είναι στον κατάλογο ψηφοφορίας της Επιτροπής. Yes, I have both. Ναι, έχω και τις δύο λίστες εδώ, οπότε μπορώ να σας πω ότι ναι, είναι στη δική μας ε, λίστα της Επιτροπής, αλλά όχι στον Σοσιαλιστό. Δεν είναι πρόβλημα της Επιτροπής. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Are we voting or not, Chairman? Okay, let's move on. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Τροπολογία 73, Πολ Μέρφη. υπέρ. Εβδομήντα τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 25 ασυγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 75 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αφέτ η 7 της αφέτ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 76 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 29 του εισηγητή και πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 30 υπέρ, 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αφέτη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην 78 τροπολογία υπέρ κατά αποχές 78 78 Πολ Μέρφυ επαναλάβουμε 78 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 79 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η ΑΦΕΤ 10 υπέρ ΑΦΕΤ 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την ΑΦΕΤ 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Λυπούμε, αλλά εγκρίθηκε. Η 80. Τροπολογία 80. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 82 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35, 35, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε άφετ 11 όχι καταπίπτει αυτή η 36 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην 38. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Άφετ 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 86 υπέρ 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έτσι δεν είναι ας ελέγξουμε ψηφίζουμε την 86 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία 86 άρχεται η ψηφοφορία The vote... πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε πράγματι Άφετ 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Άφετ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 88 τοπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αφετ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 89, 89 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αφετ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Άφετ 18 υπέρ κατά αποχές. Άφετ 18 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές. 90, 90. Η 19 κατέπεσε, η 19. Τροπολογία 90 λοιπόν. Ας επαναλάβουμε. Τροπολογία 90. Paul Murphy. διαγραφή τροπολογία. Διαγραφής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 43 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 91 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αφετήκος 20 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε να ελέγξουμε εντάξει άφετη 20 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε παρότι υπεψήφισα εγώ. Παρόλα αυτά απορριφθήκε. Ε, we Ψηφίζουμε τώρα την ΑΦΕΤ 21 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε άφετ 22 υπέρ κατά απορρίφθηκε τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε άφετ 23 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ΑΦΕΤ 23 άρχεται η ψηφοφορία And the πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα η ισοψηφία απορρίφθηκε απορρίφθηκε ΑΦΕΤ 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Σε τμήματα ξεχωριστή ψηφοφορία στο άρθρο 14 παράγραφο 3 εδάφιο 3 του εισηγητού φυσικά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε άφετ όχι η 49 τροπολογία 49 λοιπόν με προφορική τροποποίηση δεν υπάρχει κάποια ένσταση αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση λοιπόν έχετε στα χαρτοφυλάκια στους φακέλους την προφορική τροποποίηση ψηφίζουμε τη 49 λοιπόν όπως τροποποιείται προφορικά υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 50 και τροπολογία 26 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Παρατήματα. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 52. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε σκεπτικά αιτιολογικές σκέψεις σε τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε άφετ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε να ελέγξουμε ψηφίζουμε λοιπόν την 7 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία την 7 του εισηγητή άρχεται πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε τώρα τροπολογία 57. Εντάξει, όχι, η 8. Υπέρ τη 8. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 59 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Αφετ 3. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε Άφετ 3. Δεν κατέπεσε. Η Άφετ 3 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Άφετ 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε λοιπόν την ΑΦΕ 4. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is... Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε λοιπόν. Εντάξει. Και τώρα τροπολογία 11. Με προφορική τροποποίηση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για την προφορική. Όχι. Ψηφίζουμε την 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Αφετ. Όχι. Καταπίπτει. 61 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 12 υπέρ δεν κατέπεσε έτσι η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 63 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Άφετ 6 καταπίπτει, καταπίπτει 64 τώρα υπέρ. Α, το ίδιο, καταπίπτει και αυτή. 15 πάει και αυτή. 15 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 16 και 65. 16 και 65 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 66 τώρα υπέρ 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τελική ψηφοφορία τώρα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ And πέρας ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα εγκρίθηκε με 20 ψήφους υπέρ, μία κατά δύο αποχές. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα έχουμε το ψήφισμα, νομοθετικό ψήφισμα, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε γι' αυτό, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα με ίδιο αποτέλεσμα 20 ψήφοι υπέρ, μία ε, εναντίον, δύο αποχές. Τι θα κάνουμε τώρα. Είτε θα πάμε στην Ολομέλεια για ψήφιση, για ψηφοφορία ή θα περάσει άμεσα για τον άτυπο τριμερή διάλογο στις διαβουλεύσεις. Ποια είναι η πρόταση σχετικά του εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων για την υποστήριξη των γενικών ιδεών και προσέγγισης αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να ζητήσω την εντολή να περάσουμε στον άτυπο τριμερή διάλογο στις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για να καταφέρουμε να πετύχουμε έναν αποδεκτό συμβιβασμό πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Εγώ προσωπικά όλο και περισσότερο είμαι κατά του να εμπλεκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο χωρίς να έχουμε κάποια έγκριση σε σχέση με την Ολομέλεια και πολιτική συζήτηση και έγκριση όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας σε σχέση με την Ολομέλεια ξεπερνάμε έτσι ένα σημαντικό τμήμα της νομοθετικής διαδικασίας αν κάνουμε αυτό. Εγώ θα καταψηφίσω την πρότασή σας. Θα την θέσω σε ψηφοφορία φυσικά, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε τη διαδικασία, την νομοθετική, τη νομική σε σχέση με αυτές τις διαργασίες. Θα πρέπει να ζητήσουμε η Ολομέλεια να εγγράψει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη το δυνατόν ταχύτερο ώστε να μην με παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ψήφισης εδώ και της Ολομέλειας. Υπό τον όρο ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δηλαδή να έχουμε σύντομα μια συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια, εγώ θα είμαι σίγουρα κατά των διαπραγματεύσεων σε σχέση με αυτά τα θέματα, προτού έχουμε εντολή από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου δυνατότητα συζητήσεων και δυνατότητα των κοινοβουλευτικών ομάδων να καταθέσουν τροπολογίε στην Ολομέλεια. Διότι τίνουμε να ξεχνάμε ότι οι κοινοβουλευτικέ ομάδε, οι πολιτικέ ομάδε έχουν την εξουσία να θέτουν περαιτέρω τροπολογίε στην Ολομέλεια. Αν περάσουμε αμέσω στην τριμερή διαπραγμάτευση, σε τριμερή διάλογο με αποτέλεσμα αυτό το οποίο ψηφίσαμε εδώ εμεί σήμερα, θα μπορούσε, α το πω έτσι, να εκλειφθεί ω περιφρόνηση της Ολομέλειας των νέων τροπολογιών που θα ε, ψηφίζονται εκεί. Θα άλλαζαν έτσι λοιπόν, να το πω έτσι, οι κατευθύνσεις. Το θέτω υπό εξέταση. Ψηφίζουμε λοιπόν. Εγώ θα καταψηφίσω. Και εφ' εξής θα εμένω και θα επιμένω ότι θα πρέπει πρώτα να περνάμε στην Ολομέλεια. Να έχουμε εντολή από την Ολομέλεια να υπάρχει δυνατότητα οι κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες να θέτουν τροπολογίες αν επιθυμούν και αποφασίζουν έτσι, να διεξάγεται πολιτικού χαρακτήρα συζήτηση εκεί και υστερότερα μόνο να έχουμε όχι σε σχέση με την το νομοθετικό ψήφισμα στην Ολομέλεια για την πρώτη ε, ανάγνωση. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται εντολή για διαπραγμάτευση και όχι χωρίς να λαμβάνονται αυτά υπόψη. Δεν θα ήταν αυτό σωστό αν περιφρονούσαμε τη διαδικασία της Ολομέλειας. Τούτων λεχθέντων ψηφίζουμε την πρόταση του εισηγητή να περάσουμε αμέσως σε άτυπες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Εγώ καταψηφίζω, θα προσθεθεί η ψήφος μου στις ψήφους κατά. Τέλος ψηφοφορίας. Και πράγματι απορρίφθηκε λοιπόν. Εντάξει, απορρίφθηκε η πρότασή σας. Εσείς παρακαλώ. Oui, Monsieur le Κύριε Πρόεδρε, είπατε την προσωπική σας άποψη για τη διαδικασία. Νομίζω όμως ότι χρήζει μιας πραγματικής συζήτησης, γιατί για ορισμένα θέματα θα ήταν άκρος ενδιαφέρον να ξεκινήσουν γρήγορα διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εκφράσατε εσείς την άποψή σας, απόλυτα θεμητή, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να το συζητήσουμε και ο καθένας να εκφράσει τη δική του άποψη για το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα δόγμα οριστικό. Υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις ε, στις διάφορες επιτροπές και παραλαμβάνω, ορισμένες φορές ε, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν πάρα πολύ γρήγορα οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα ήταν καλό να κάνουμε μια συζήτηση. Πρόεδρο, συμφωνώ μαζί σας ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια πλήρη συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά κάποια συζήτηση έχει ήδη γίνει. Εγώ θα είχα δώσει το λόγο σε οποιονδήποτε μου το είχε ζητήσει. Ο Παύλ Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα μπορούσε πράγματι να υπάρξουν ε, θέματα που θα είχε νόημα να προχωρήσουμε ομαλά στις διαπραγματεύσεις και γρήγορα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αλλά αυτό θα πρέπει να θεωρείται εξαίρεση, διότι εν γέννη πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ισχυρή εντολή από την Ολομέλεια. Διότι έτσι η θέση μας στις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν θα ισχυροποιηθεί. Κατά δεύτερον, συμφωνώ ότι σε ορισμένες περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσει. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι ο κανόνα. Ευχαριστώ. Uh, η κυρία Κφίστχου του Ρόμπολ. Πρέπει να πω στον συνάδελφο Ζαντό ότι όλοι μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μα ε, ψηφίζοντα. υπέρ ή κατά. Ε, δεν είναι ανάγκη να γίνει συζήτηση και να χαθεί χρόνο. Μπορούμε να πούμε ναι ή όχι. Ο κύριος Αντώ προφανώς είπε ναι, εμείς ήμασταν κατά της πρότασης του συναδέλφου Κάζακ και το ίδιο ακριβώς θα γίνει και για το επόμενο θέμα. Θα ψηφίσουμε εδώ, στην Επιτροπή μας, για μια ακόμη φορά. Ο Πρόεδρος. Ωραία, το σημειώσαμε αυτό. Ίσως να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής μας ε, το θέμα αυτό προς θα έχουμε ένα γενικό κανόνα. Βέβαια πάντα χωρούν εξαιρέσεις στους κανόνες, αλλά μετά από την εμπειρία μου, διότι έχω προεδρεύσει όλων των τριμέρων διαλόγων, νιώθω ότι είναι πιο ισχυρή η θέση μας εάν έχουμε την ε, ψηφό της Ολομέλειας. Ξέρετε ότι θέλω πάρα πολύ να προεδρεύω των διαπραγματεύσεων Σίγουρα βέβαια αφήνω τον κάστοτε συγκεκριτή να ηγηθεί της διαδικασίας αλλά και ως παρατηρητής και ως εισηγητής επίσης σε πολλά θέματα έχω καταλάβει ότι η θέση μας είναι πολύ ισχυρότερη όταν έχουμε πίσω μας την ψήφο της Ολομέλης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι μετά την ψήφο στην Επιτροπή να περιμένουμε δύο μήνες να πάει το θέμα στην Ολομέλη. Αυτό ναι, δεν είναι σωστό και πρέπει να αλλάξει. νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να φέρουμε το θέμα προς ψήφιση των ολομέλεια το συντομότερο δυνατόν. Επομένως θα πιέσουμε τη διάσκεψη των Προέδρων και βέβαια κυριότερα τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου να αλλάξουν τις διαδικασίες και πρακτικές για να μην υπάρχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. μεταξύ της εδώ ψηφοφορίας και της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Λοιπόν, ψηφίσαμε και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεύτερη ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας. Έκθεση της Χωσέφα Αντρές για την εξωτερική διάσταση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Γνωμοδότηση είναι για την Επιτροπή ΠΕΣ Αλίας που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ας ψηφίσουμε λοιπόν την γνωμοδότηση με τις τροπολογίες. Ξεκινάμε τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ελέγχει, θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 3, μάλιστα, άρχεται η ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορία. Εγώ σας είπα ότι θα καταψηφίσω, άρα καταψηφίστηκε για τα 10 προς 10. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε την τροπολογία 8. Άρχεται ψηφοφορία. Εγώ θα ψηφίσω κατά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 περ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία του σχέδιου νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγώ ψηφίζω υπέρ. And it was Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στη Χωσέφα. Εδώ λοιπόν λήγουν ε, οι σημερινές μας ψηφοφορίες και περνάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Στο σημείο, συγγνώμη, 30. Okay. Well, let's, uh, folks, let's settle down. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ να έχω την προσοχή σας. Could you stop your conversations? Could you sit down? Παρακαλώ σταματήστε τα παραθυράκια και τα πηγαδάκια μάλλον και καθίστε. people standing. Να μην βλέπω ορθίους παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τώρα στο σήμερα 30 ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριο Κοζίρο Σιοζίρι. warm, warm welcome to you and to your um, σας καλωσορίζουμε πως και την ομάδα σας. Μετά από την μεγάλη καταστροφή στην Ιαπωνία, θα ήθελα να τη φόρο τιμής εκ μέρους της Επιτροπής μας στον τρόπο με τον οποίο εσείς αντιμετωπίσατε την φαβερή αυτή ναι. καταστροφή. Μετά το τσουνάμι και το σεισμό, μάλλον μετά το σεισμό και το τσουνάμι, ξεκίνησαν τεράστιες προσπάθειες ανοικοδόμησης, αποκατάστασης και επειδή έχω πάει και έχω δει τι γίνεται επί τόπου, μπορώ να σας πω ότι πραγματικά υπάρχει μια πανεθνική δέσμευση από όλους τους Ιάπωνες. Η Ιαπωνία γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί και επιδεικνύει αλληλεγγύη προς την Ιαπωνία, βοηθά όσο μπορεί. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Επιτροπή μας. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η επίσκεψή σας, γιατί υπάρχει μια διερευνητική ε, άσκηση η οποία έγινε για να δούμε κατά πόσο πληρούνται οι προποθέσει για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει για μια μελλοντική εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία έχουν προοδεύσει τα πράγματα και ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να ολοκληρωθούν. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε την άποψή σας και για αυτό το θέμα αλλά και για το όλο φάσμα των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Σας δίνουμε πολύ μεγάλη χαρά τον λόγο κύριε Πρέσβη. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια. Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για τις ε, εμπορικές σχέσεις Ιαπωνίας ΕΕ, χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές σχέσεις παγκόσμια. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια έκθεση υποεξέλιξη σε αυτό το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή σε σχέση με την αλληλεγγύη για την ανοικοδόμηση ένα χρόνο μετά το μεγάλο σεισμό στην Ανατολική Ιαπωνία. Δεν θα ξεχάσουμε την αλληλεγγύη που έδειξαν οι ευρωπαϊκοί λαοί χωρίς προηγούμενο αλληλεγγύη, σε αυτή την χωρίς προηγούμενο καταστροφή της Ιαπωνίας. Δράτω με τις ευκαιρίες για άλλη μια φορά για να εκφράσω τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη σε όλους σας και πράγματι στην Ευρώπη που προσπαθεί η Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση χρέους σε αυτό το σημείο είχε αγοράσει ομόλογα του ESFF η Ιαπωνία και έτσι δείχνουμε την αλληλεγγύη μας και η Ιαπωνία έχει προαναγγείλει την συμμετοχή της σε ύψος 60 δις δολαρίων και ενθαρρύνει και άλλους να ακολουθήσει το παράδειγμά μας παρόλες τις, ε, τα, τα προβλήματα τα οποία αγωνίζεται να ξεπεράσει η Ιαπωνία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ίδια. Θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας έναντι της Ευρώπης. Όπως εσείς μας συνδράματε, εμάς τους Ιάπωνες, έτσι και εμείς να σας βοηθήσουμε. Μετά από αυτή την καταστροφή μάθαμε το ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την πρόοδό μας. Παρότι είναι πολύ δύσκολη και είναι πραγματικά πολύ αντίξωη η κατάσταση και διανοίγεται έτσι η οδός για την ανάκαμψη και αναδιάρθρωση, ανοικοδόμηση της ε, Ιαπωνίας και με την βοήθεια εκτός. Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία διαβούλευσης για την ε, δι... και στις δύο όχθες του ειρηνικού συνεργασία και διανοίγεται και η δυνατότητα μεταξύ ΕΕ Ιαπωνίας και με την αναγνώριση που δείχνεται από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2011 για μια νέα εμπορική πολιτική της Ευρώπης με τον στόχο της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020 αυτή η έκθεση λέει σαφώς ότι ε, το εμπόριο συνεισφέρει στις, ε, ε, στην ανταγωνιστικότητα και συνεισφέρει με σημαντικά προτερήματα υπέρ των καταναλωτών. Θέλουμε μέσα από αυτή τη νέα σχέση να πούμε ότι ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα με τα συμπεράσματα της έκθεσής σας. Σήμερα θέλω να επαναλάβω και να τονίσω τους στόχους μας και τη στεναρότητά μας, τη δέσμευσή μας, να έχουμε μια νέα φιλόδοξη τέτοια σχέση με την ΕΕ. Οι στόχοι που ακολουθούνται μέσω της ε, ε σύμβασης αυτής, της συμφωνίας αυτής, είναι η αναζωγόνηση των οικονομιών μας οι αποφάσεις ε, της κυβέρνησής μας όσον αφορά την πολιτική για μια σφαιρική εμπορική εταιρική σχέση μέσω της κυβέρνησής μας είμαστε στεναρά αποφασισμένοι και δεσμευμένοι να είμαστε προπομπή για ένα νέο μέλλον μέσα από αυτή την οικονομική εμπορική εταιρική σχέση. Και η Ιαπωνία και η ΕΕ αντιμετωπίζουν δύο κοινέ προκλήσεις, την δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών σχέσεων και ε, αυξημένων επενδύσεων. Δεύτερον, για τη νέα αυτή οικονομική και παγκόσμια διάσταση πρέπει ΕΕ και η Ιαπωνία να αναλάβουν ρόλο πρωτοπόρων. Εμείς ε, σε σχέση με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με τις υφιστάμενες αυτές εταιρικές ε, συμφωνίες και με την Κίνα, μια εταιρική τέτοια συμφωνία καθιστά την Ιαπωνία ιδανικό εταίρο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δίνοντας συνέχεια σε αυτούς τους δύο στόχους θα πρέπει να επιτύχουμε την ανοικοδόμηση, την, ε, ενίσχυση των οικονομιών μας που πρέπει να είναι καινοτόμες, ανταγωνιστικές και αιφόρες. βιώσιμες στο μέγιστο ενθυμούμενοι πάντα ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία ήταν πάντα πρωτοπόροι στην παγκόσμια σκηνή προς ε, την κατεύθυνση αυτή. Υπό το φως της σημερινής κατάστασης σε σχέση με τον γύρο της Ντόχα, η Ιαπωνία και ΕΕ θα πρέπει να οδηγήσουμε και να θέσουμε κατευθύνσεις σε άλλες χώρες, ε, δίνοντας το καλό παράδειγμα, υιοθετώντα τις βέλτιστες προδιαγραφές για τις οικονομικές συμφωνίες, ε, όντας παγκόσμιοι πρωτοπόροι για να πετύχουμε αυτούς τους ίστατους, ιστερότερους στόχους, εμείς από πλευρά της Ιαπωνίας σοβαρά εμπλεκόμεθα σε, με σοβαρό τρόπο σε ρυθμιστικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ως τμήμα της δικής μας μεταρρύθμισης για την ανάπτυξη. Αυτό ήταν αυτό το οποίο επανειλημμένα εξέθεσε και εξέθεται ο Πρωθυπουργό μας. Δηλαδή να αναζωογονηθούν αυτές οι προσπάθειες και αυτή η προσπάθεια είναι πραγματικά σημαντική για τις μεταρρυθμίσεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Νόντα είναι υπεύθυνο και επικεφαλής αυτών των διαδικασιών. Και υπήρξε και συνάντηση στο, στη στρογγυλή τράπεζα ΕΕ Ιαπωνίας. Οι συστάσεις ζητούν να επιταχυνθούν οι ρυθμοί και οι διεργασίες ε, υπό το φως ε, της ε, επιτυχούς ολοκλήρωσης σε αυτό το εγχείρημα το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συστάσεις κάνουμε λόγο για το εύρος το πλαίσιο και το επίπεδο φιλοδοξιών που είναι ιδιαίτερα υψηλό προσεγγίζουμε την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών τώρα και πιστεύουμε ότι η θετική αυτή πρωτοβουλία θα στέψει με επιτυχία τις διαβουλεύσεις και το διάλογο αυτό. Οι διαπραγματεύσεις ε, θα ξεκινήσουν και καταδεικνύουμε σαφώς την προθυμία μας και την ικανότητά μας να ρυθμίσουμε, να ε, θέσουμε εντάξει τις ρυθμιστικές διατάξεις που ενδιαφέρεται η Ευρώπη να επιτύχει αναφέρατε την κυβερνητική ε, μονάδα αναζωογόνησης, αναφέρθηκε αυτή που καταβάλει προσπάθειες σε σχέση με τα ειδικά αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα υπάρξει συνεισφορά για την αναζωογόνηση με συζητήσεις σε αυτή τη μονάδα. Από πέρυσι οι αρχές στην Ιαπωνία έχουν ήδη αναλάβει συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα σε συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά για παράδειγμα τις πρόσθετες ουσίες στα τρόφιμα και άλλα θέματα. Σε αυτή την έκθεση του Απριλίου που κατατέθηκε με προτάσεις ε, του τι θα έπρεπε να γίνει σε σχέση με τον εξοπλισμό ε, των ε, διαφορετικών ηλεκτρονικών συσκευών, επίσης για την πρόοδο όσον αφορά εξοπλισμό με συσκευές διαφόρων οχημάτων, προϊόντα ε, και σε σχέση με την ε, κυβερνητική προμή, τις κυβερνητικές προμήθειες δημιουργήσαμε ένα one-stop shop για την παροχή πληροφοριών που ξεπερνά τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ που έχουμε αναλάβει. Υλοποιώντας ε, τις ε, υποχρεώσεις μας, αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε και άλλα θέματα μη δασμολογικά, ώστε να υπάρξουν διευρυμένες δυνατότητες για τις ε, προμήθειες και συμβάσεις. Από πέρσι ο διάλογος μεταξύ των βιομηχανιών της Ιαπωνίας και της Ευρώπης προάχθηκε με ενεργό τρόπο με στρογγυλές τράπεζες και με την Νιπών, και την, τις επιχειρηματικές οργανώσεις της Ευρώπης για θέματα αυτοκινητοβιομηχανιών, πληροφοριών, επικοινωνίας των πληροφοριών, κλωστοϊφαντουργίας, ε, ασφάλειας χημικών προϊόντων, ιατρικού εξοπλισμού, φαρμακευτικών προϊόντων υπήρξαν αντίστοιχοι διάλογοι που αναπτύχθηκαν ε, μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας. Επίσης διάλογος για τον τομέα τον σιδηροδρομικό που ε, διαοργανώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Όλες, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες διαλόγων όχι μόνο θα ενισχύσουν την εμπορική μας σχέση αλλά θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες μας με επιτυχή τρόπο. Έχουμε και το scoping exercise με τις επαφές αυτές και χωρίς αμφιβολία μπορούμε να πούμε ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές θα αντανακλώνται όλες οι προσπάθειες. Τα πιο σημαντικά που μπορούν να επιτευχθούν είναι να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα για τις επιχειρήσεις και για τις βιομηχανίες της Ευρώπης και της Ιαπωνίας οι σχέσεις ΕΕ και Ιαπωνίας ε, θα διευρύνουν περαιτέρω τις δυνατότητες για επενδύσεις και για την εξαγωγή ε, προϊόντων. Πριν από 30 χρόνια, ως νέος διπλωμάτης τότε, εργαζόμουν στην Ιαπωνική αποστολή στις ευρωπαϊκές κοινότητες, όπως τις αποκαλούσαμε τότε. Υπήρχαν έντονες εμπορικές τριβές τότε, όπως για παράδειγμα στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα και στα ηλεκτρονικά. Και συχνά τονιζόταν και τονίστηκε ότι θα ήταν αναγκαίο να ενισχυθούν οι σχέσεις μας, οι σχέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρώπης. Μετά από τρεις δεκαετίες ολόκληρες επανήλθα στις Βρυξέλλες ως πρέσβης πλέον της Ιαπωνίας ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου αποστολή έγκυται στο να διευρύνουμε τις σχέσεις μας στο επίπεδο εκείνο το οποίο είναι ευκταίο όσον αφορά να είμαστε, για να είμαστε υπεύθυνοι παγκόσμιοι ηγέτες. Θεωρώ ότι η ολοκλήρωση της EPA είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος θα έπρεπε να δραχθούμε της ευκαιρίας και να μην χάσουμε την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται. Ευχαριστώ για την προσοχή. Uh, well, let's open the... Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, έχουμε αποφασίσει πριν από κάποιους μήνες ε, ότι θα θεσπίσουμε εντός της Επιτροπής μας μια, μια μόνιμη ε, ομάδα παρακολούθησης για, τους, για κάθε έναν από τους πιο σημαντικούς μας εμπορικούς εταίρους. Προφανώς ένας εξ αυτών είναι η Ιαπωνία. Ο μόνιμος εισηγητής για την μόνιμη αυτή ομάδα είναι ο Μέτιν Καζάκ από την ομάδα Άλντε, στον οποίο θα δώσω το λόγο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Με την, έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κύριε Πρέζοη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τη δήλωσή σας. Με χαρά άκουσα την ισχυρή δέσμευση που μας κάνατε ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και να επιτύχετε τα αμοιβαία επιθυμητά αποτελέσματα και ενδεχομένω και την έναρξη δηλαδή των διαπραγματεύσεων για την οικονομική εταιρική συμφωνία μεταξύ Ένωση και Ιαπωνία. Όπω θα θυμάστε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για τι εμπορικέ σχέσει μεταξύ Ένωση και Ιαπωνία στι 4 Μαου του περασμένου έτους. Λίγο μετά την υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματο, η διάσκεψη κορυφής Ένωση Ιαπωνία ξεκίνησε την διαδικασία διαπραγματεύσεων για μια βαθιά και συνολική εμπορική συμφωνία ε, και ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα scoping. Εγώ προσωπικά είμαι ένθερμος υποστηριχτής αυτής της πρωτοβουλίας. Ωστόσο, εξ αρχής το Κοινοβούλιο επίσης υπογράμμισε πως η Ιαπωνία θα πρέπει να αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για την άρση των μη δοσμολογικών ε, φραγμών καθώς και τα εμπόδια στις ε, Ιαπωνέζικες δημόσιες συμβάσεις πριν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας ε, έχει μείνει πίσω σε σχέση με αυτό με άλλους εμπορικούς μας Σύμφωνα με ακαδημαϊκές μελέτες όπως η οικονομική μελέτη της Κομμεχαής, αυτό οφείλεται βασικά στην αρνητική επίπτωση των ε, Ιαπωνικών μη, μη δεσμολογικών φραγμών. Γι' αυτό και με απογοήτευσε που άκουσα ότι το σκόπινγκ δεν μπορεί να τελειώσει ε, το Μάρτιο γιατί ε, κρεμούν ζητήματα για τις γεωγραφικές ενδείξεις καθώς ε, και τα MTB και τις δημόσιες συμβάσεις. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πάρει θέση στις διαπραγματεύσεις στην Ολομέλεια του Ιουνίου μάλλον αν μπορέσουμε να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα μέχρι τότε και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την έναρξη μιας ε, ε, εμπορική συμφωνία Ένωση Ιαπωνία όταν θα ανοίξουν και οι δημόσιε συμβάσει. Θα πρέπει να έχουμε παρκή ωφέλη σε αντάλλαγμα για να αιτιολογήσουμε την μείωση των δασμών για τα αυτοκίνητα και τα ηλεκτρονικά τις ηλεκτρονικές συσκευές. Έπειτα χρειαζόμαστε ένα δεσμευτικό μηχανισμό στη μελλοντική με, συμφωνία, ώστε να μην υπάρξουν νέοι ε, μη δεσμολογικοί φραγμοί στην Ιαπωνία. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει ε, μέγα δυναμικό και πιστεύω πως μια τέτοια συμφωνία είναι η σωστή προσέγγιση για να τονωθεί η αγορά τόσο της Ιαπωνίας όσο και της Ένωσης. Όμως πιστικά αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την άρση των ε, εμπορικών ε, φραγμών πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και ελπίζω Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι τον Βάιο θα μπορέσουμε να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα για να έχουμε και ισχυρότερες θέσεις και να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, the other members of the monitoring group uh, are uh, shadows uh, from... Και τώρα θα πάρουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες ομάδες. Για Ροσλάβ Βαλέσα από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα πω πολλά αλλά νομίζω ότι η απογοήτευση είναι η λέξη κλειδί. Γιατί ακόμα μια χρονιά πέρασε και δεν έχουμε και πολλά να επιδείξουμε. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος ε, του Μαΐου να έχουμε κάποια, ένα οδικό χάρτη για να δούμε ποια, ποια εμπόδια ακόμα πρέπει να ξεπεραστούν, όπως τα μη δασμολογικά, η μη δασμολογική φραγμή και όλα αυτά για τα οποία ζητάμε από τον περασμένο Μάρτιο. Εάν δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς προσπαθούμε να επιτύχουμε με αυτές τις διαπραγματεύσεις, θα καταλήξουμε σε ακόμα μια χαμένη χρονιά και θα βρισκόμαστε στην ίδια θέση πάλι. Ελπίζω λοιπόν ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις παρά ερωτήσεις. Και εγώ είμαι μέλος αυτής της ομάδας ε, εποπτείας, καθώς είμαι και μέλος... Θα πρέπει να σας πω εγώ πως εγώ δεν είμαι απογοητευμένος. λόγω της καθυστέρησης αυτής της ε, προσπάθειας. Γιατί από την αρχή ξέρω ότι δεν θα ήταν εύκολο. Δεν ξέρουμε πόσο πολύ επιθυμεί η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις διασφαλίσεις ότι η, Ευρωπα... η Ιαπωνική πλευρά θα μπορέσει να δεσμευτεί όσον αφορά του μη δασμολογικού φραγμού και εφόσον μετέβηνε και δύο φορέ και έχω μελετήσει την Ιαπωνική κατάσταση, ξέρω ότι πολλέ αντιστάσει θα πρέπει να ξεπεραστούν στην Ιαπωνία ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Πολύ δύσκολα ζητήματα λοιπόν που χρειάζονται χρόνο και πολιτική βούληση για να επιληθούν. Υπάρχει πολιτική βούληση στην Ιαπωνία πιστεύω, αλλά οι προκλήσεις είναι τεράστιες ώστε να και απαιτούν μάλλον χρόνο και πολλή προσπάθεια. Ελπίζω πως τελικά θα επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. αλλά κατανοώ επίσης γιατί δεν έχουμε προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο θα περίμεναν μερικοί. Ας αφήσουμε λοιπόν χώρο και στα δύο μέρη να μελετήσουν την κατάσταση, να δουν μήπως υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω πως ο πιο εύκολος τρόπος ε, για να αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις είναι όταν η ε, διαπραγματεύσεις χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει μια τέτοια δραστηριότητα. Θα πρέπει να περιμένουμε να οριμάσει η κατάσταση. το... Από ό,τι κατάλαβα στην ιαπωνική πλευρά ασχολούνται και έχουν δεσμευτεί πολιτικά για μια οικονομική εμπορική συμφωνία και με τον ειρηνικό κεφάλαιο και με την υπερακυρινική ε, εταιρική συνεργασία είναι μεγάλες προκλήσεις και είναι ένα μεγάλο σοκ για την ιαπωνική οικονομία αυτό άνοιγμα που, που αναζητούμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Μια διμερής εμπορική συμφωνία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται δυο για να λειτουργήσει. Δυο εταίρους, όπως και το ταγκό. Mm. Τα πράγματα προχωρούν. Δεν, υπάρχει, δεν, δεν έχουν τελματωθεί συζητήσεις, αν και προχωρούν αργά, αν και αργά σταθερά. ακούσουμε και την Κομισιόνα για να δούμε ποια είναι η άποψη της ευρωπαϊκής πλευράς. Η Κομισιόν χρειάζεται την στήριξη του Κοινοβουλίου και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η θέση της Κομισιόν. όταν έχουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να δείξουμε στους συνομολητές μας μια πολύ ισχυρή οικονομική, ε, πολιτική θέση. Συγγνώμη. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει ξεκάθαρη θέση και πιστεύω πως η Κομισιόν συμφωνεί. Ας δούμε λοιπόν τη γνώμη του κύριου Ζάραντιλ. Ευχαριστώ πολύ. Ξοχώτες, κύριε Πρέσβη. Κυρίε και κύριοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία αυτή είναι προ αμοιβαίο όφελο, προ όφελο δηλαδή και των δύο πλευρών και συμφωνώ και με τι ανησυχίε αλλά και με τι ελπίδε που εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι όπω οι κύριοι Καζά και Βαλένσα για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα λεπτό ζήτημα που αποτελεί κομμάτι της μέσιας διάταξης, δηλαδή ο τομέας των δημόσιων συμβάσεων, κυρίως για την αεροπορία και το σιδηρόδρομο. Ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να μπορέσουν να ανταγωνιστούν και σε αυτό τον τομέα να έχουν πρόσβαση στις συμβάσεις αυτές. Θα ήθελα λοιπόν η Ιαπωνική πλευρά να μας δώσει κάποιες ενδείξεις πώς έχουν τα πράγματα, τι θέση έχουν αυτή τη στιγμή και τι εξελίξεις θα μπορούσαμε να αναμένουμε στο μέλλον. για να δημιουργηθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για να δούμε πώς, πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε. Παραλαμβάνω ότι δεν θέλω να ε, με διακατέχει απελπισία, αλλά η αισιοδοξία σε σχέση με την ε, κατάσταση και την πρώτη των διαπραγματεύσεων. Ο Μπεν Λάγκε τώρα έχει το λόγο από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας εδώ και για τα την σαφή σας τοποθέτηση ότι αυτή η συμφωνία είναι προς το κοινό συμφέρον ενίσχυσης των εμπορικών μας σχέσεων. Αυτό το υπογραμμίζω και το προσυπογράφω απόλυτα. Όμως φυσικά ήδη αναφέρατε και ένα κρίσιμο πεδίο στο οποίο, το οποίο πρέπει να έχουμε ενώπιόν μας, δηλαδή τα θέματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ξέρετε κύριε Πρέσβη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι η βιομηχανία πυρήνας στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει και δυσκολίες σε αυτή τη συγκυρία που αντιμετωπίζει. Στον προβληματισμό μας για μια τέτοια εμπορική συμφωνία πρέπει ακριβώς να μεριμνήσουμε τα συμφέροντα της αυτοκινητοβιομηχανίας αυτής να αντανακλώνται όσον αφορά την Ευρώπη. Και αν δει κανείς αυτό το τμήμα, τρεις τομείς, τρεις άξονες υπάρχουν, κύριε Πρέσβιο, που μπορεί κανείς να ρωτήσει και να δει. Είναι αποδεκτό τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταίρων να μην λαμβάνονται υπόψη εμπορικά όπως πρόκειται, όταν πρόκειται για το θέμα πιο φιλοπεριβαλλοντικών αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία Ιαπωνικά οχήματα με Ιαπωνικές δοκιμασίες προτιμώνται και δεν υπάρχει αντιστοιχία σε σχέση με τις δικές μας διεργασίες. Δεύτερον, το θέμα φορολόγησης των αυτοκινήτων. Και εδώ φαίνεται η φορολόγηση στην Ιαπωνία να μην αντιμετωπίζει θέμα δασμολογικών ε, ε, προσκομμάτων και εμποδίων. Και το τρίτο, αν δούμε το άνοιγμα της αγοράς, με την πώληση αυτοκινήτων δεν επιλύονται όλα τα προβλήματα αυτόματα. Υπάρχει το θέμα των συνεργείων και ανταλλακτικών και τα λοιπά και εμπόρων. Και αν δούμε ότι σε σχέση με την νομοθεσία όσον αφορά τον αποκλεισμό εμπόρων, εκπροσώπων και συνεργείων πρέπει αρκετά και πολλά πράγματα να γίνουν για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να συνάψουμε μια τέτοια εμπορική συμφωνία. Ίσως μπορείτε να μας εκφράσετε, να μας εκθέσετε κάποιες σκέψεις σας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Και τέλος, λέει ο Πρόεδρος, να σας πω ότι ικανοποιούμαστε ιδιαίτερα να έχουμε τον Πρόεδρο ανάμεσά μας της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Ιαπωνία τον συνάδελφο κύριο Φανμπάλεν. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας και ευχαριστώ για την επίσκεψή σας και τη συμμετοχή σας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Και φυσικά μπορείτε να παρέμβετε για να μας εκθέσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το θέμα αυτό. E Ευχαριστώ πολύ. Ως αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ιαπωνία θα συνέλθουμε με τους εταίρους μας της Ιαπωνικής Δίαιτας τον Μάιο να δούμε ποια εμπόδια και δυσκολίες υπάρχουν και πρέπει να ξεπεράσουμε. Μπορούμε να έχουμε έτσι μια θετική ολοκλήρωση του scoping exercise. Ευχαριστώ. Who is the Commission? εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αντώνιο Παρέντα, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΡΕΙΝΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Ούτε κύριε Πρέσβη, Ισιογύρη, αγαπητοί βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία και για τα σχόλια. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η συζήτηση αυτή, διότι Ελπίζουμε και από ό,τι φαίνεται πράγματι, ερχόμαστε στην τελευταία φάση των συνομιλιών για την ε, προπαρασκευή της έκθεσης αυτής ε, διερεύνησης μετά αυτό το scoping exercise. Ε, βέβαια, είναι δύσκολο να προβλέψουμε ακριβώς πώς θα εξελίξουν τα πράγματα και εμείς το ανέφερε και ο Ιάπωνας πρέσβης. Λάβαμε πρόσφατα μια πολύ σημαντική απόφαση. We think of a sea change in the attitude that the Japanese government has. Uh, που σηματοδοτεί μάλλον ε, μια αλλαγή πλεύσης από την Ιαπωνική κυβέρνηση γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα που για πολλά ε, χρόνια ε, παρακόλιαν τις διμερείς απορικές μας σχέσεις. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά του GRU. αλλά θα επαναλάβω ε, ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η ανάλυση του έργου αυτής της ομάδας ε, συνεχίζεται και θα είναι και στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα έχουμε με τους ε, Ιάπωνες συναδέλφους μας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το θέμα, μάλλον τα θέματα, είναι ιδιαίτερα τεχνικά θέματα τα οποία συζητώνται στο επίπεδο του GRU και γι' αυτό θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν θα εισέλθω σε λεπτομέρειε, δεν μπορώ να σα κάνω μια πλήρη εκτίμηση, γιατί ακόμα βρισκόμαστε σε φάση εξέταση όλων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, για τι διαπραγματεύσει και για την ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η Κομισιόν ε, μελετά όλα τα πράγματα. Είδαμε να επιβεβαιώνονται και οι δύο στόχοι και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε αν ε, η Ιαπωνία μπορεί να δείξει ότι υπάρχει κρίσιμη μάζα μη εμπορικών φραγμών τα οποία, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξαλειφθούν και περιμένουμε επίσης επίλυση ζητημάτων που είναι πολύ σημαντικά για μας ε, παραδείγματο χάρη δημόσια συμβάση, ιδίω στον συνδρομικό τομέα. Ο στόχος μας είναι η, ε, το αίσιο πέρας των συνομιλιών και δεν μας ενδιαφέρει τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο να υπάρξει αίσιο πέρας παραλαμβάνω. Είναι και ο Επίτροπος Δεχούχτ μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια με τον Επίτροπο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ε, πολύ λογικό να του ζητήσω αφού είναι εδώ να μα μιλήσει και αυτό για τι εμπορικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, Ιαπωνία. επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Να πω ότι συμφωνώ βέβαια απόλυτα με αυτό που είπε ο εκπρόσωπος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ. Μπαρέντι. Αλλά στο πολιτικό μέτωπο θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμεί στην Κομισιόν και η ΓΔΤ Trade θέλουμε σίγουρα μια συμφωνία με την Ιαπωνία δεν ακολουθιεργούμε σε καμία περίπτωση, δεν ακολουθούμε μια παρελκυστική τακτική. Απ' την άλλη πλευρά, προτού ξεκινήσουμε τελικά τις διαπραγματεύσεις, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι θα έχουν ένα αίσιο αποτέλεσμα, ένα αίσιο πέρας. Άρα πρέπει προηγουμένως να συμφωνήσουμε με την ε, Ιαπωνική κυβέρνηση για μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τους NTBs, τους μη εμπορικούς ε, φραγμούς. Αναλύουμε τις προτάσεις που εκ πρώτης όψης φαίνεται να συνιστούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Η Ιαπωνική κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός και το καλωσορίζουμε αυτό. Βέβαια, όλα αυτά είναι προτάσεις και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ιαπωνική κυβέρνηση να δείξει στην πράξη ότι κάνει πράξη αυτά τα οποία έχει προτείνει. Καλή την πίστη. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα πράγματα ε, στην πράξη. Είναι όμως ένα να βγούμε προς τα εμπρός και θέλω να ευχαριστήσω τους ε, Ιάπωνες ομολόγους για τις προτάσεις τους. Εργαζόμαστε λοιπόν με πολύ ταχύς ρυθμούς και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να είναι όλα έτοιμα για να μπορέσουμε να έχουμε και μια διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας στην οποία διάσκεψη κορυφής θα έχουμε πλέον μόνο την επιλογή. Ναι ή όχι. Δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Δεν μπορούν να είναι ανοιχτέ όλε οι δυνατότητε. Ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο και στο μέλλον τη διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ιαπων Πρέσβης έχει πάλι το λόγο. Για να απαντήσει στις ερωτήσεις και τα σχόλια των ε, βουλευτών της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι, αυτό το scoping exercise ε, το υιοθετούμε και προσεγγίζουμε την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος. Μέσω των πολύ σοβαρών προσπαθειών μας σε αυτό το scoping exercise μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα κοινή κατανόησης και προσέγγισης και έτσι θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε υψηλό επίπεδο scoping και φιλόδοξο, μεγάλης φιλοδοξίας επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πιστεύουμε. Σε διαφορετικά θέματα που αναφέρθηκαν, αυτοκινητοβιομηχανία, σιδηρόδρομοι, αεροπλάνα κτλ. κτλ. Ανέφερα προηγούμενα στην παρέμβασή μου το πιο σημαντικό για μας, το οποίο έγκυται στις διαπραγματεύσεις EPA, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον για επιχειρήσεις και για τις ε, ιαπωνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα είναι θετικό Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις απόψεις σας και όπως προανέφερα στον λόγο που εξεφώνησα ήδη υπάρχει καλό κλίμα συζητήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και της Ευρώπης. Προσβλέπουμε λοιπόν σημαντικά στο να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα scoping και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ πολύ πρέσβη πολύ καρποφόρα, πολύ γόνιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση εξάλλου. Φυσικά το ότι προσήλθατε είναι θετικό και είσαστε και πρόσδεκτος. Κυρίε και κύριοι, ας περάσουμε στο σημείο 31 τώρα. Έχουμε και την Επιτροπή, τον Επίτροπο για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική για το εμπόριο για μας την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αυτό αποτελεί τμήμα των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον διαρθρωμένο διάλογο, δομημένο διάλογο μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και με ψήφισμα από την Ευρωβουλή μας. Νομίζω αυτό το στόχο θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση να εμπλακείτε σε αυτές τις συζητήσεις προπαρασκευαστικά προ... ετοιμάζοντας αυτό το διάλογο ώστε ως συνομοθέτες να μπορέσουμε να δράσουμε και όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας να μπορέσουμε να δράσουμε πλήρως. Κύριε Επίτροπε, είσαστε τακτικά ε, επίτροπος που προσφωνεί την Επιτροπή μας και μας επισκέπτεστε και αυτό δείχνει την καρποφόρα και σε βάθος συνεργασία μεταξύ μας και μεταξύ ημών. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Ανάλογα με το πόσο μετρά κανείς δεν έχουμε μόνο 3,5 χρόνια που είμαστε στην ε, μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά από την ε, μεγάλη ύφεση, την ε, Επιπλέον είμαστε, μάλλον επικρατούν διάφορα οι παράγοντες στην παγκόσμια οικονομία που υποβαθμίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και η εμπορική πολιτική βρίσκεται στην καρδιά για της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Το να ανοίξουμε νέες αγορές είναι ο φτηνότερος τρόπος για να κινητοποιηθεί η ανάπτυξη που χρειαζόμαστε. Και όπως ξέρουμε, Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη θα γίνει εκτός ε, των σύνορων της Ένωσης και άρα χρειαζόμαστε αποτελεσματική ε, εμπορική πολιτική ώστε να επανέλθει κάποια από αυτήν την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι αυτή η επιστρατηγική μπορεί να είναι ποτέ η Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ καλός έμπορος. Είμαστε ο μεγαλύτερο εξαγωγέας και εισαγωγέας μεταποιημένων αγαθών. 20% του συνόλου μεγαλύτερος ε, άμεσος επενδυτής ε, εκτός Ένωσης παραμένουμε επίσης και αποδέκτης ξένων επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά μας για το εμπόριο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη ε, είναι κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης και γι' αυτό έχουμε μια επιτακτική ευθύνη απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή να δώσουμε νέες ευκαιρίες στην οικονομία μας να αναπτυχθεί. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, οι συζητήσεις όπως η σημερινή είναι πολύ σημαντικές. Ελπίζω πως θα συμφωνήσετε πως μπορέσαμε να έχουμε τακτικές εις βάθος συζητήσεις για ένα μέγα φάσμα θεμάτων κλειδιών. Αλλά τώρα έχουμε μια στιγμή για να ε, κάνουμε μια αναθεώρηση. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι είμαστε στο ίμιση της εντολής του Κοινοβουλίου και του μου εντολή ω επιτρόπου. Αν θέλουμε να σηματοδοτήσουμε τη διαφορά για τα θέματα όλα αυτά, θα πρέπει να αρπάξουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Και ελπίζω πως θα μπορέσουμε επικοδομητικά να ενεργήσουμε μαζί για την δημιουργία θέσεων απασχόληση και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας με την ίδια ένταση όπως και στο πρώτο ήμιση της θητείας μας. Πρόκειται για μια περίοδο που δικαιωμάσαμε νέες διαδικασίες ε, μέσω της συνθήκης τη Αβώνας. Δεν ήταν όλα ομαλά. Γίνανε συζητήσεις για τις, ε, ε, θέματα όπως η επιτροπολογία που πήραν πολύ καιρό, περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Ελπίζω λοιπόν πως θα κλείσουν οι διαδικασίες για όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε άσχημα όσον αφορά το επιτεύγματά μας για τη διαφάνεια και ε, μάλιστα μπορεί να παρουσιαστούν και νέα διαδικαστικά ζητήματα, για να, αλλά πάντοτε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε χωρίς εμπόδια. Η διαδικασία ε, εκμάθησης ε, ήταν απότομα ανηφορική και για τις δύο πλευρές. Για να εν συντομία την Συμφωνία Άκτα. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν επίση πόσο πολύ είμαι ε, προσιλωμένο στη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε ε, συζητήσει το Άκτα εδώ και τρία χρόνια και θα το συζητήσουμε ακόμα. Μέχρι χτε η βασική επίκριση ήταν ότι η Άκτα είναι αόριστη. Τώρα ακούω για συγκεκριμένα θέματα που θεωρείται ότι λείπουν ή που πρέπει να αποσαφινιστούν στη Συμφωνία έτσι όπω έχει σήμερα. Ας το συζητήσουμε λοιπόν. Αυτό που αντιπροσωπεύει η άκτα όσον αφορά τις θέσεις στην ανάπτυξη στην για την Ευρώπη χρειάζεται, αξίζει να συζητηθεί πλήρως, δημοκρατικά. Θα ήθελα να σας δώσω μια γενική εικόνα των βασικών ζητημάτων πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση υπό τον τίτλο «Εμπορικές διαπραγματεύσεις, σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους και θέματα πολιτικής». Πρώτον, για τις διαπραγματεύσεις. Προχωρούμε προς ε, τους μακροπρόθεσμους στόχους μας ε, για την επίτευξη συμφωνίας με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Η Σιγκαπούρη μπορεί να είναι η πρώτο μου αποτέλεσμα. Ε, είναι ένα σημαντικό εμπορικό εταίρος της περιοχής και όχι μόνο γιατί 9.000 ευρωπαϊκές εταιρείες χρησιμοποιούν ως κέντρο την Σιγκαπούρη, αλλά και επειδή έχουμε διαπραγματευτεί φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Επίση, είναι στο κέντρο μιας περιοχής που είναι φυσικός μας εταίρος. Όταν ε, συναντήθηκα με τον Υπουργό Λίν τον περασμένο μήνα στην Πνομ κάναμε σημαντική πρόοδο και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Τώρα, η συμφωνία με τη Μαλαισία μπορεί να είναι η δεύτερη. Έχουν γίνει πρόοδοι, αλλά υπάρχουν ακόμα προκλήσεις ε, για τα αγαθά όπως ε, τα αυτοκίνητα και υπηρεσίες αλλά και οι δημόσιες συμβάσεις. Στο Βιετνάμ, τρίτος ε, τέρος μας ε, ε, ΑΣΕΑΝ, θα συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό Χουάν στα τέλη του, του μήνα. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων για την συμφωνία, την εμπορική ελεύθερων συναλλαγών. Επίσης έχουμε προχωρήσει στην οικονομική συμφωνία με τον Καναδά. Φιλοδοξία και των δύο πλευρών να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις το 2012. Γνωρίζουμε ήδη πως τέτοιου είδους συμφωνίες ε, φέρουν σημαντικά ωφέλη. 99% των δασμών επί αγαθών θα καταργηθούν μέσα σε 7 χρόνια. Θα σημάνει επίσης σημαντικά ανοίγματα για τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις από τις διάφορες επαρχές του Καναδά, για τις διάφορες επαρχές του Καναδά. Ωστόσο παραμένουν δύσκολα ζητήματα που ως επίλυση, όπως ε, για παράδειγμα η πρόοδος όσον αφορά την πρέση για τα αγαθά, όπου έχουμε σκαλώσει στους κανόνες προέλευσης. Επίσης αναμένεται απόφαση ε, μεσοπρόθεσμα για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και του πλαισίου υπό το οποίο θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα ήδη είπα. Έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας για το ποια ακριβώ είναι οι νέε προτάσεις της Ιαπωνίας και πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές. Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω την, τις οικονομική οικονομικής συνεργασίας, εταιρική σχέσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, κατάλληλη ε, περίοδος για τις διαπραγματεύσεις. Η... Το 2012 θα είναι κρίσιμο για να επιληθεί η κατάσταση των ενδιάμεσων ε, ε, οικονομικών εταιρικών συμφωνιών που έχουν εγκριθεί το 2007 αλλά δεν έχουν επικυρωθεί από την αφρικανική ε, πλευρά. Για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να διατηρηθεί η όθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει σε αυτά υιοθετώντα την προτινόμενη τροπολογία για, ε, για τον κανονισμό πρόσβασης στην αγορά. Η στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα στέρεο και ε, νομικό πλαίσιο για ε, τους εταίρους μας συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων μας και διαπραγματευτών μας στην Αφρική. Το κάνουμε αυτό με τις χώρες Ανατολικής Αφρικής. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να προχωρήσει για τις συμφωνίες που ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε συμφωνίες με την Κολομβία, Περού, Κεντρική Αμερική. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω τις παρατηρήσεις μας πως αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν σημαντικό οικονομικό δυναμικό και για τις δύο πλευρές. Επίσης πληρούν απόλυτα τις προσδοκίες της Ένωσης και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι επιτυχής η κατάσταση εκεί και θα πρέπει πλέον να προχωρήσουμε. Έχουμε επίσης τις σχέσεις μας με τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω όλους εδώ γιατί θα συζητηθούν περαιτέρω σήμερα, αλλά είναι σημαντική η δουλειά που θα κάνουμε στου επόμενου μήνε για την Κίνα, γιατί είναι η χώρα που αντιπροσωπεύει τι μεγαλύτερε ευκαιρίε και τι μεγαλύτερε προκλήσει για τι πολιτικέ μα. Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενη εξαγωγική μα αγορά και αντούμπαλιν είμαστε εμεί για αυτήν. Όμω έχουμε και με ένα μακρύ κατάλογο προβλημάτων με την Κίνα και γι' αυτό θα συνεχίσουμε στεναρά να ενεργούμε στον ΠΟΕ για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. The Commission's procurement initiative is not... Η πρωτοβουλία των δημοσίων συμβάσεων δεν αφορά την Κίνα, αλλά θα την αφορά αν την εγκρίνεται ως ένα μέσο για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να εξασφαλίσουμε το καλύτερη πρόσβαση των εταιριών μας στις ξένες αγορές. Επίσης, δουλεύουμε για μια θετική ατζέντα για τη συνεργασία και την καινοτομία, πράγμα το οποίο είναι βασικό για την ατζέντα της Κίνας. Αν μπορέσουμε γρήγορα να μπούμε με ισότιμους όρους, οι οικονομικές προοπτικές μπορούν να είναι πολλά υποσχόμενες. Οι επενδύσεις είναι ένα στο τομέα, αλλά θα επανέλθω στο θέμα των επενδύσεων αργότερα. Τώρα, δεν μπορώ παρά να τονίσω επίσης τη σημασία της προσχώρηση της Ρωσία στον ΠΟΕ μετά από 18 χρόνια διαπραγματεύσεων. Αυτή η εξέλιξη μας δίνει νέα μέσα για να ασχοληθούμε, να αντιμετωπίσουμε τα προστατευτικά μέσα των Ρώσων. Για παράδειγμα, καταστήσαμε σαφέ ότι η απαγόρευση των εξαγωγών ζών των ζώων από την Ευρώπη ε, ε, των εισαγωγών μάλλον από την Ευρώπη είναι απαράδεκτη. Επίσης ε, θα, πρέπει, θα έχει να αντιμετωπίσει με το που θα προσχωρήσει το ΠΟΕ ρύθμιση διαφορών και σχετικά πάνελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σταθερά να επιμείνει στο ότι μια νέα συμφωνία με τη Ρωσία χωρίς εμπόριο και συμφωνίες για την ενέργεια δεν θα είχε νόημα. Αλλά για μας είναι σημαντικός ο στόχος αυτός για τη διάσκεψη κορυφής Ένωσης Ρωσίας τον Ιούνιο. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε πλήρη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Όμως δεν πρέπει να τρέχουμε αυτά πάτες ότι, ε, ότι πρόκειται για ένα πολύ μακρόπνο πρόγραμμα. Λόγω της ε, Τελωνιακής με το Καζακστάν και τη Λευκορωσία δεν μπορεί πλέον να διαπραγματεύεται μόνη της. Τώρα, για τις συγκεκριμένες πολιτικές σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε για τις επενδύσεις. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς ε, ταραχτήκατε με τα όσα έκανε η Αργεντινή για τη Ρέψολ. Πολύ ατυχές βήμα από την ε, προοπτική του αργεντινικού λαού, του οποίου η κυβέρνηση διακυβεύει θέτει σε κίνδυνο μάλλον την μελλοντική του ε, ευημερία ήταν ιδιαίτερα είναι ιδιαίτερα ατυχής η κατάσταση και για την Ισπανία και κοιτάμε, εξετάζουμε ό,τι δυνατότητα έχουμε στη διαθεσή μας για να απαντήσουμε μια σειρά αδικαιολόγητων ε, προστατευτικών μέτρων που ελήφθησαν και εισήχθησαν πρόσφατα από την Αργεντινή. Όμως, αυτή η κατάσταση μας θυμίζει το πόσο σημαντικό είναι να κινηθούμε γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα μέσα που χρειαζόμαστε για την επενδυτική μας, τις επενδυτικές μας πολιτικές υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις διμερείς επενδυτικές συνθήκες των κρατών μελών, προχωρούμε. Η πρόσφατη συνένεση που πετύχαμε το Συμβούλιο είναι πολλά υποσχόμενη. Εννοείται ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να διευκολύνει το τελικό συμβαστικό κείμενο και ελπίζω πως αυτό θα γίνει σύντομα ώστε να υπάρξει νομική ε, βεβαιότητα για τους επενδυτές μας. Επίσης προχωρούμε με τις νέες διαπραγματεύσεις περί επενδύσεων. Προωθούμε ε, διαπραγματεύσεις ε, προστασίας των επενδύσεων με τις νότιες μεσογειακές χώρες, τη Σιγκαπούρη, τον Καναδά και την η Ιαπωνία και επίσης θα διαπραγματευτούμε την προστασία των επενδύσεων με άλλους εταίρους ε, ΑΣΕΑΝ. Έχουμε επίσης παρακινήσει την παροτρύνη την Κίνα να προχωρήσει προς ε, την ε, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά με την, την, και ήδη κάνουμε περισσότερες προετοιμασίες γιατί κάτι τέτοιο θα είναι πολύ σημαντικό βήμα. Σύντομα επίσης θα λάβετε πρόταση σε σχέση με την οικονομική ευθύνη του επενδυτή για την ε, επίλυση ε, διαφορών ε, κατόπιν των αποφάσεων που ελήφθησαν τον Απρίλιο. Είναι πολύ σημαντικό τμήμα της αρχιτεκτονικής μιας ευρωπαϊκής επενδυτικής πολιτικής. Σύντομα θα λάβετε και πρόταση για έναν κανονισμό για την επιβολή των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων μετά από τις ε, διμερείς και περιφερειακές ρυθμίσεις διαφορών στον ΠΟΕ. Ε, θα μπορούμε να σκεφτούμε και αντίπεινα για να προστατέψουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, μέσα στο χρόνο θα εξετάσουμε τις δυνατότητες εξοχρονισμού των ε, εμπορικών μέσων ε, άμυνας που ε, θα έχουμε και αυτά θα τα δείτε στο 2013 στο Κοινοβούλιο. Μιλήσαμε επίσης για διαφάνεια με τους εταίρους μας και έχουμε θα κάνουμε μια μεγάλη διάσκεψη στα τέλη Μαΐου. Η τελευταία προσπάθεια σε αυτό το τομέα έχει αποτύχει, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και θα αποφύγουμε την επανάληψη αυτό. Να ζητούμε σύγκληση απόψεων για ένα ισορροπημένο πακέτο, όπως απειλέ αντιπίνων κατά τη ευρωπαϊκή βιομηχανία, διαφάνεια και επιβολή. Όπως μπορείτε να δείτε, στόχος μας είναι να εστιάσουμε στα πρακτικά προβλήματα των πραγματικών επιχειρήσεων και να μην προβούμε σε ιδεολογική συζήτηση για το κατά πόσο τα μέσα ή αυτά που χρησιμοποιούμε είναι εξαιρετικά φιλελεύθερα, προστατευτικά ή κάτι άλλο. Αυτά εμπίπτουν στην ατζέντα που σας ανέφερα και προηγουμένως που στόχο έχει τη συμβολή στο εμπόριο, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αλλά έχω την εντύπωση, κοιτώντας την ατζέντα σας κάθε φορά που έρχομαι εδώ, και αυτό συμβαίνει συχνά, ότι η Επιτροπή σας είναι μια από τις πιο πολυάσχολες στο Κοινοβούλιο. Σε, αυτές τις ε, περιόδους, σε αυτή την περίοδο κρίσης αυτό που, δεν έχουμε μπροστά, που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο που σημαντική δουλειά, πολλή δουλειά αλλά και σημαντική δουλειά. Και όπως είπα και στην αρχή η δουλειά είναι πολύ σημαντική ώστε να εξασφαλίσουμε πως η Ευρώπη θα μείνει στο μονοπάτι της ευημερία ε, ενώπιον της μέσα σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Εγώ έρχομαι εδώ σε στενή συνεργασία θέλω να εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα καταφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε δεν κάνατε μόνο έναν απολογισμό και μια επισκόπηση των ε, συζητημάτων ε, που μας απασχολούν αυτόν τον καιρό, αλλά κάνετε και κάποιες ε, ανακοινώσεις για τις επενδύσεις και κάποιους εμπορικούς μηχανισμούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση ακούγοντας εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. ΕΛΚ καταρχάς, ποιος θα εκπροσωπήσει το ΕΛΚ. Εσείς, η κυρία Κβίστοφουτ Ρόβολ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ ενώπιόν μας και ευχαριστώ που, ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Επίτροπε επαναλαμβάνει η ομιλήτρια και ευχαριστώ που διαρκώς μεριμνάτε να είσαστε σε φάση, σε επαφή και διάλογο μαζί μας και τουλάχιστον υπάρχουν τόσο πολλά διαφορετικά θέματα που υπάρχουν, βρίσκονται υπό εξέταση που έτσι συμπυκνωμένα όταν τα ακούμε από εσάς πραγματικά μας εκπλήσει. Υπάρχουν τόσα πράγματα που θα έπρεπε να μας ε, απασχολήσουν. Εκείνο όμως το οποίο προσέχω ιδιαίτερα και παρατηρώ σε αυτά τα οποία λέτε είναι ένα μόνιμο σημείο. Όλο και περισσότερο κινούμαστε στο επίπεδο διμερών συμφωνιών και συνθήκων. Λάθος δεν είναι αυτό και όταν κάτι δεν λειτουργεί πολυμερός κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε εντάξει διμερός πολύ καλά. Η ερώτησή μου στοχεύει όμως προς το εξή. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση ας το πω έτσι του πολυμερούς πλαισίου. Πολύ ωραία είναι να γίνει μέλος του ΠΟΕ η Ρωσία αλλά αν δεν θα σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο όταν δεν θα υπάρχει ισομερής αντιμετώπιση σε σχέση με όλους. Ναι μεν χαιρόμαστε την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ αλλά δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Εντάξει, δεύτερη ερώτηση. Όλες οι διαπραγματεύσεις αυτές που γίνονται με την Κεντρική και Νότια Αμερική υπάρχει, τουλάχιστον εγώ αυτό μπορώ να περιγράψω από τη δική μου περιφέρεια, όλο και περισσότερο αντίσταση. Αντίσταση από κάθε μίκιο ενώσεις συλλόγους πολιτών που πιστεύουν ότι πολύ άνισα είναι όλα αυτά και στο τέλος τέλος τι υποστηρίζουμε υποστηρίζουμε δικτατορικά καθεστώτα ή μη δημοκρατικά καθεστώτα και κυρίως στο τέλος τέλος τι κάνουμε δομές και διαθρώσεις υπονομεύουμε και καταστρέφουμε σε αυτές τις χώρες με τη δράση μας πρώτον ερώτηση κατά πόσον έχουμε προχωρήσει σε αυτά. Ολοκληρώνεται, τερματίζεται αυτό και βλέπετε κάτι εσείς υπό το πρίσμα σας να έχει αλλάξει σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια νέα κίνηση, κάποια αλλαγή. Και μία ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω σε σχέση με τη Συμφωνία Άκτα για την πνευματική ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα. Εχθές κιόλας είχαμε την, πρέσβη, την πρέσβυρα εδώ όσον αφορά τις ΙΠΑ ε, και συζητήσαμε ανοιχτά και ειλικρινά μαζί της. Έχω την εντύπωση και αυτό ξεχωριστά από τη δική μου άποψη αν είμαι υπέρ ή κατά εγώ όλων αυτών έχω την εντύπωση που αποκόμισα ότι το συνολικό πλαίσιο παίρνει τέτοια μορφή που εντάξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι ε, κάτι που λαμβάνεται υπόψη, όμως οι άλλοι σταυρώνουν τα χέρια τους και περιμένουν και αναμένουν να δουν τις εξελίξεις. Ποια είναι η δική σας ε, εξέλιξη αντικειμενικά για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από αυτή την υπογραφή, αν προσυπεγράφεται και ενεκρίνεται το η άκτα τι πιστεύετε εσείς και μια εξειδικευμένη συγκεκριμένη ερώτηση. Διαρκώς έχουμε διαπραγματεύσεις και επαφές με την Τουρκία. Εντάξει, τώρα από την κλωστοϊφαντουργία έχουμε ακούσει για δραματικά παράπονα και προσφυγές όσον αφορά δασμολόγια, δασμολογικές επιβαρύνσεις ε, όσον αφορά την Τουρκία που οξύνουν την κατάσταση όλο και περισσότερο. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτά τα θέματα και τις διαπραγματεύσεις και κυρίως όταν υπάρχουν τέτοιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ως συμβάντα πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Όλα είναι ωραία ως θέματα αρχών, αλλά όταν έχουμε εξειδικευμένα θέματα ως προβλήματα, τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μεν Λάγκε τώρα από τους σοσιαλιστές. Κύριος Λάγκε, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, σας ευχαριστώ και σας πολύ για τον διαρκή διάλογο που καλλιεργείτε μαζί μας με την Επιτροπή μας. Δύο θεματικά πλέγματα. Πρώτον, και το ερώτημα του μέλλοντος για το μέλλον του ΠΟΕ. Δεν το ε, εστιάσατε ιδιαίτερα. Μιλήσατε για όλο το φάσμα της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που φυσικά σε πολλούς τομείς συνεπάγεται και διμερείς διαπραγματεύσεις. Εντάξει, όταν όμως έχουμε πολλές διμερείς ε, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που συνάπτουμε που δεν αφορούν μόνο θέματα δασμών και δασμολογίων αλλά και αφορούν και θέματα ουσιώδη νομοθεσίας των χωρών εταίρων. Τι γίνεται με το εμπόριο. Αυτές οι διαφορετικές δομές ε, δεν αποτελούν ένα στενότερο πλαίσιο και μια επιδίνωση και υπονόμευση του πολυμερούς πλαισίου διεθνώς. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα πώς εκτιμάτε τις μελλοντικές προοπτικές. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει μια δυνατότητα αυτό το στένεμα του ε, εύρους, του φάσματος ε, να το αποφύγουμε και να είμαστε πολυμερέστεροι. Δεύτερο θέμα, Trade Defense Instruments με ξέπληξε κάπως ε, για το ότι αυτό έχει πάλι επανεγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Καλό είναι βέβαια να έχουμε ένα δημόσιο ανοιχτό διάλογο που θα διοργανώνεται έτσι και θα γίνει η ακρόαση στις 10 Μαΐου, αλλά να εξειδικευθεί περισσότερο. Πού βλέπετε ακριβώς τις προκλήσεις ή τις ε, αναγκαιότητες βελτιώσεων έναντι του σημερινού, της σημερινής κατάστασης. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ. Μέρος ομάδας Άλντε. Έχει το λόγο ο κύριος ε, Κάζακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εντάξει, με ακούτε. Με ακούτε. Ακούγεται η Γερμηνία. Yeah единство в многообразието, все пак. Това е девизът на Европейския съюз. А, господин комисар. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω και προσωπικά αλλά και εκ μέρου της ομάδας μου για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που κάνατε, την επισκόπηση αυτή των διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με τις ε, διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη και με τους εμπορικούς μας εταίρους και με τρίτους. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να στεφθούμε με επιτυχία όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το τονίσατε και εσείς πάνω από μία φορά, δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχουν για την ε, υπέρβαση αυτής της οικονομικής κρίσης και την διάνοιξη νέων επενδυτικών και εμπορικών ε, οριζόντων για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σιγκαπούρη, Μαλαισία. Νομίζω ότι τις πρόλες συναντήθηκε η ομάδα παρακολούθησε τις χώρες αυτές. Έχουμε μεγάλη πρόοδο. Είναι ξεκάθαρο ότι και ως προς τις δύο αυτές χώρες και ως προς την Ιαπωνία υπάρχουν κάποια εμπόδια παρόλα αυτά, κυρίως αφορούν τους κανόνες προέλευσης και τις δημόσιες συμβάσεις. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, εφόσον υπάρχει κάτι τέτοιο, για το πότε περιμένετε να υπερπηδηθούν όλες αυτές οι δυσκολίες. Αυτό ήταν το πρώτο μου σχόλιο. Δεύτερο. Γνωρίζετε ότι υπάρχει προτινόμενη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων, GPA. Υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας από την Κομισιόν, το οποίο επικεντρώνεται σε μέτρα προστατευτισμού απέναντι σε τρίτες χώρες, άνοιγμα ή κλείσιμο ε, των κρατικών μας προμηθειών ε, προς ε, τρίτες χώρες ανάλογα με τις δράσεις που λαμβάνουν αμοιβαίως οι χώρες αυτές. Εξ όσων γνωρίζω δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη για το σύνολο όλων αυτών. Παραδείγματος χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο άκρος φιλελεύθερα σκέπτεται. Άλλα κράτη-μέλη όμως επιμένουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως η αρχή της πλήρους αμοιβαιότητας. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε τη διαφωνία που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών μας. Πώς θα προασπίσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση αποφεύγοντας ταυτόχρονα αντιπαραγωγικές ε, δράσεις, δηλαδή το να αποκόψουμε την πρόσβαση στις αγορές μας ε, για εταίρους που είναι παρόλα αυτά σημαντικοί για εμάς. ECR, ποιος θα λάβει το λόγο, ο Γιάν ε, Ζάχραντιλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και τον Επίτροπο. που πάντοτε μας παρουσιάζει πολύ πρακτικές προσεγγίσεις, ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Είπατε ότι η Επιτροπή μας είναι μια από τις πλέον πολύ άσχολες. Νόμιζα θα πείτε ότι είναι και μια από τις σοφότερες επιτροπές σε ό,τι αφορά την μέση διάταξη και την ε, υλοποίησή της. Σας ευχαριστώ πάντως για την πολύ πλήρη αυτή παρουσίαση. Θα ήθελα να σχολιάσω τρία σημεία. I know. You, you, you, you can't do this. Um, thank you for mentioning... Σας ευχαριστώ γιατί αναφερθήκατε για μια ακόμη φορά στις EPA, δηλαδή τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Η Επιτροπή μας πολύ πρόσφατα επισκέφθηκε την Ανατολική Αφρική. Και πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν και άκρο θετική εμπειρία μας. Είχαμε δηλαδή ενίοτε την εντύπωση ότι κάποια μέλη της διοίκησης όλων ή ορισμένων χωρών από αυτή την περιοχή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί να προχωρήσουν και για συγκεκριμένους, πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν περισσότερα από εσάς για το πώς αξιολογείτε εσείς αυτή την κατάσταση και ποιες προοπτικές βλέπετε για περαιτέρω ανάπτυξη ενός πλαισίου με την Ανατολική και την ε, Νότια Αφρική σε σχέση με τις ε, συμφωνίες ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Βιετνάμ θα ήθελα επίσης κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, αν έχετε. Φαίνεται να έχει σημειωθεί αρκετά ικανοποιητική πρόοδος μέχρι στιγμής. Και σας θέτω το συγκεκριμένο αυτό ερώτημα, όχι τόσο ως εκπρόσωπος μιας συγκεκριμένης πολιτικής ομάδας, αλλά ως μόνιμος εισηγητής για τη συμφωνία αυτή εξ ονόματος της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Αν είναι δυνατόν λοιπόν θα σας παρακαλούσα να αναφέρετε κάποια ισχυρά και κάποια αδύναμα σημεία αυτής της ε, διαδικασίας. Α, και κάτι ενδιαφέρον, δεν είναι και ίσως πάρα πολύ γνωστό, η μεγαλύτερη βιετναμέζικη κοινότητα από με σχετικούς όρους, σε σχέση δηλαδή με τον συνολικό ρυθμό κατοίκων στην Ευρώπη, ζει στην Τσεχία, τη χώρα μου. Η σχετικά μεγαλύτερη βιετναμέζικη μειονότητα στην Ευρώπη. Γι' αυτό με ενδιαφέρουν ακόμη περισσότερο όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις και βέβαια οι ομαλή τους ε, υλοποίηση και ολοκλήρωση. Οι συμφωνίες τώρα ελεύθερων συναλλαγών με Κολομβία και Περού, σαν να τέρμονη μοιάζει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια αίσια ευτυχής ολοκλήρωση. για τη συγκεκριμένη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών, νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ακριβώς η προσέγγιση που μας εκθέσατε στην αρχή της ομιλίας σας. Αυτή δηλαδή η πρακτική και ρεαλιστική προσέγγιση. Ελπίζω να συμφωνείτε και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο William Dartmouth. Mm. Έχω να κάνω κάποιε ερωτήσει. Εμπορική Συμφωνία Ένωση Ινδία. Μπορείτε να μας πείτε ποια πρόοδο έχει γίνει, αν έχει γίνει. Και επίση εν γέννη, δεν θέλω να σας βάλω σε δύσκολη θέση, αλλά σα έγραψα στις 21 Μαρτίου, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Ο βοηθό μου με διαβεβαιώνει πως είναι στάνταρ καθυστέρηση ένα μήνα σε, σε αυτό το είδο τη λογραφίες. Υπήρξε μια έκθεση στις ε, Βρετανικές εφημερίδες για ότι four uh, in the treaty. Έγινε αναφορά λοιπόν για τον ε, τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται η μετανάστευση και ότι mode for στην συνθήκη. Δεν κατάλαβα. Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι Πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσει Ένωση Ινδία. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι. ότι στις Βρετανικές εφημερίδες υπήρξαν αναφορές ότι ως τμήμα της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας θα θα είναι μια ρήτρα που θα σχετίζεται με τη μετανάστευση από εκεί. Αυτά τα είπαν οι Βρετανικέ εφημερίδε και εγώ σα έχω στείλει σχετική επιστολή και έχω κάνει και ερώτηση σε προηγούμενη ευκαιρία που ήσασταν εδώ. Η απάντησή σα ήταν πάρα πολύ, πολύ ξεκάθαρη. Αλλά ίσω οι Βρετανικέ εφημερίδε θα πρέπει να διορθωθούν, γιατί δεν λένε πάντοτε την αλήθεια, απαραίτητο. Uh, ε, no. okay. no, no, but not yet. other members. Uh, uh, για σύντομη ερώτηση, τώρα θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ο Ντέιβιντ Μάρτιν πρώτα. Και μετά η Σιλβάνα Κοχμέριν. Τρεις ερωτήσεις. Αλλά σας καθυσυχάζω, είναι όλες τις σύντομες. Άκτα. Τι έχουμε να πούμε για το άκτα. Τι να συζητήσουμε. Είπατε ότι ήταν, παλιά λέγαμε ότι είναι αόριστη και ότι τώρα ακούτε πιο συγκεκριμένες επικρίσεις. Αλλά ακόμα και έτσι, και τι να κάνουμε για τις επικρίσεις αφού ήδη έχει εγκριθεί μια συνθήκη που έχει υπογραφεί από όλους τους εταίρους. Δεύτερον, ε, κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά. Ο ισχύων δεν έχει καταληκτήρια ημερομηνία. Είναι σαφέ ότι η Κομισιόν είναι δεσμευμένη και προσιλωμένη στην, στην ημερομηνία πρώτης πρώτου. Γιατί αποφασίσετε για αυτή την ημερομηνία και γιατί όχι 30 Ιανουαρίου, ε, ε, Ιουνίου 2014 ή 2013, γιατί η συγκεκριμένη ημερομηνία, ποιο λόγος σας οδήγησε στην θέση αυτής της ημερομηνίας. Και τρίτη και τελευταία μου ερώτηση, είναι σαφές ότι σε κάποιες από τις διαπραγματεύσεις μας Ε, είναι σαφές ότι έχουμε πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις όταν εκεί έχουμε TPP. Οι Αμερικανοί ας πούμε δεν προωθούν τα GI όταν υπάρχουν TPP. Και υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύσεις ε, αλλάζουν κατεύθυνση ε, και ότι εμείς αποδυναμωνόμαστε στις διαπραγματεύσεις. Ισχύει αυτό ή όχι. Η Κυρία Κόχμαριν, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η μία φορά τον Καναδά. Πέρσι όλοι ελπίζαμε ότι θα Ολοκληρωθεί η ΣΥΤΕΡ ε, φέτος. Ε, τώρα όλοι ξέρουμε πώς θα γίνει για τον πάει για τον επόμενο χρόνο. Ξέρουμε ότι η δεξιά και η αριστερά διαπραγματεύεται ο Καναδάς με άλλους εμπορικούς εταίρους. Τι μπορούμε να κάνουμε για να επιτεχυνθεί η διαδικασία ε, ώστε να μην χάσει τη σημασία της και το νόημά της. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο Χεντεγκάρντα Ελπίζω πως οι εμπορικές ε, πτυχές θα συμπεριληφθούν σε ε, μελέτη αντικτύπου. Και δεύτερη ερώτηση για τη Ρωσία. Εσείς υπογραμμίσατε τη σημασία της ένταξης της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. τη νέα, τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, αν δείτε ότι υπάρχει μια νέα δυναμική ε, του ΠΟΕ και της ε, προσχώρησης και για άλλες χώρες τέρους στην Ανατολική προς Ανατολάς, ποια είναι η εικόνα σας και έπειτα για τις γαλλικές ε, εκλογές. Πώς νομίζετε πως αυτές θα επηρεάσουν την εμπορική πολιτική ελευθέρων συναλλαγών της Κομισιόν. Και εγώ δύο ερωτήσεις. Πρώτον για την άκτα. Η πρώτη είναι συνταγματική φύση. αν μπορεί να ψηφιστεί ενώ το θέμα έχει παραμευθεί στο, κοινοβούλιο, ε, στο δικαστήριο. Ποια είναι η άποψη της Κομισιόν. Και έπειτα, Αν απορριφθεί η άκτα και φοβούμε πως αυτό θα γίνει, τα άλλα συμβελάμενα μέρη θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τη συμφωνία μεταξύ τους. Ποιες είναι οι ενδείξεις που έχετε. <clears throat> Έχουμε χρόνο λοιπόν, έχετε χρόνο και θα έχουμε και την κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίας. Επιλέξτε λοιπόν πώς θα μας ενημερώσετε. Μικρόφωνο παρακαλώ. Because many, uh, uh, of these... Πολλά από αυτά τα θέματα αξίζουν, όχι μόνο αξίζουν, αλλά πρέπει να τύχουν εξαντλητικής απάντησης. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά ερωτήματα διατυπώθηκαν από την κυρία Κβίστα Ρόβοτ και από τον κύριο Μπέντ Λάγκ εξάλλου για το διμερές, πολυμερές πλαίσιο του ΠΟΕ και τα λοιπά, τα συναφή αυτά θέματα. Μάλιστα, I believe, I... πιστεύω, ειλικρινά το πιστεύω, ότι είναι σφάλμα σφάλμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει στο πολυμερές επίπεδο αυτών των συμφωνιών. Πιστεύω είναι σφάλμα και θα το αναγνωρίσουμε και στο μέλλον. Αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε μόνοι μας. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως εξήγησα αρκετές φορές ενώπιον της κοινοβουλευτικής σας επιτροπής, πρόκειται για το για την αξιολόγηση που έχει κανείς, πώς βλέπει κανείς τα πράγματα, για αυτό που θα έπρεπε να στοχεύει να πετύχει όσον αφορά τον γύρο της Ντόχα. Η Ντόχα ξεκίνησε πάνω κάτω πριν από δέκα χρόνια. Στο μεσοδιάστημα ο κόσμος άλλαξε, δεν έμεινε ακίνητος. Είχαμε τις αναδυόμενες οικονομίες που εμφανίστηκαν, θέματα ανταγωνισμού και το θέμα είναι τι θα πρέπει να παραμείνει από τις ασύμμετρες αυτές σχέσεις που οδήγησαν στην Ντόχα οι ασύμμετρες σχέσεις σε σχέση με τις αναδυόμενες οικονομίες, τις ε, ανεπτυγμένες οικονομίες στις υπόλοιπες χώρες. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι ένας συμβιβασμός θα είχε νόημα να επιτευχθεί. Γι' αυτό προτείναμε να έχουμε τομεακά για τα θέματα των μηχανών, των ε, χημικών κτλ. Αλλά δεν συμφωνούν όλοι από αυτού. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς ε, προτείναμε τουλάχιστον να προσπαθούσαμε να επιλύσουμε το θέμα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, LDCs, και είμαστε σε πολύ καλή θέση, διότι δίνουμε τα πάντα εκτός από όπλα στις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στην ε, κάτω του Ισημερινού, την νότια του Ισημερινού Μεσημβρινή Αφρική και αλλού. Είναι πολύ σημαντικό όμως δεν έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις εφόλων ε, των θεμάτων. Το ίδιο και για το βαμβάκι παράδειγμα. Και όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά είναι πολύ σημαντικά αυτά. Και αν δει κανείς τις πρόσφατες ταραχές ε, όσον αφορά τη ζώνη του Βάμβακα στο Μαγρέμ δεν είναι χωρίς πολιτικές ε, επιπτώσεις και χωρίς τη σπουδαιότητά τους όλα αυτά. Η ιδέα είναι τώρα να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων. Πολύ σημαντικό αυτό. Να δημιουργηθεί μια θέση win-win, αμφωτέρωθεν προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα υιοθετήσουν ξαφνικά και θα δεχθούν αυτό ως ένα γεγονός κάτι το αναπόφευκτο θα κατανοήσετε το τι εννοώ. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό να εξεταστεί εκτός του συνολικού πλαισίου. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το προσεγγίσουμε και να το επιλύσουμε με μια φιλόδοξη συμφωνία για το μέσο, για το εμπόριο να, το να μπορούσαμε σε σχέση με την Τόχα να προχωρήσουμε, αλλά χρειάζεται το πολιτικό θάρρος να ε, συναθριστούν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε προς μια τέτοιου είδους συμφωνία. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να συμβεί αυτό, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε πρόοδο πολυμερός, στην αυθεντική έννοια σημασιολογικά της έννοιας πολυμερός διότι ακόμα και εκτός ε, MFN ε, αν κάτι δεν είναι αυτού του χαρακτήρα και είναι διμερούς ε, πλαισίου πώς μπορεί κανείς να πετύχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν και υπάρχει μια παρανόηση ουσιώδης. Όμως θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε, να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το πλαίσιο. Η κυρία Κρίστα Ρόβοτ επίσης έθεσε ένα ερώτημα σε σχέση με την Νότια Αμερική. Από ό,τι κατάλαβα από την ερώτησή σας κυρία Κρίστα Ρόβοτ, εννοείται Κολομβία, Περού, έτσι δεν είναι. Είδα, ήδη είπα επανειλημμένα στη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρηθεί μια καλή συμφωνία. Είναι ένα καλό πλαίσιο αυτό Έχουμε πολλές διασφαλίσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου σε σχέση με αυτές τις χώρες. Αν μόνο συνάπτουμε συμφωνίες με εταίρους όπου δεν μπορούν να υπάρχουν οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις, ε, τότε θα μπορέσει να διευκολυνθεί η, η δουλειά μας. Όταν έχουμε καταλάβει, καταβάλει κάθε προσπάθεια να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία και ελπίζω ότι και το Ευρωκοινοβούλιο θα το αξιολογήσει, θα προχωρήσουμε έτσι. Μετά υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την άκτα. Θα επανέλθω όμως υστερότερα στο τέλος ε, της παρέμβασής μου σε αυτό. Ας το αφήσουμε αυτό λοιπόν τελευταίο στην ε, διευθέτησή του. Για την Τουρκία μάλιστα υπάρχουν προβλήματα σίγουρα και πήγα και στην Τουρκία. Πότε ήταν 5-6 μήνες πριν, εν πάση περιπτώσει, η Τελωνιακή Ένωση δεν λειτουργεί καλά με τους Τούρκους και τους το είπαμε των Τούρκων αυτό το πράγμα. Και εκείνοι δυσαρεστούνται. Και ένας από τους λόγους είναι ότι όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και δεν, απο... δεν είμαστε απόλυτα μέρος των εμπλεκόμενων μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε υποβάλει προτάσεις ώστε να είμαστε πιο στενά συνδεδεμένοι μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Μέχρι στιγμή δεν υπήρξε όμως κάποια ανταπόκριση, αντίδραση από τους Τούρκους επ' αυτού. Από την άλλη πλευρά έχουμε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μαζί τους όπου πιστεύω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ενώπιον του ΠΟΕ. Μέχρι στιγμή δεν υπήρξε ένα πάνελ διότι δεν καταλήξαμε σε προσφυγή, διότι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με τις καλές μας προθέσεις να επιλύσουμε τα προβλήματα. Αλλά πρέπει και η Τουρκία να σημειώσει πρόοδο για να επιτευχθεί αυτό. Η Τελωνιακή Ένωση είναι μια συμφωνία, εντάξει. Και οι δύο συμβαλόμενοι εταίροι πρέπει να έρθουν στο ύψος των απαιτήσεων και περιστάσεων. Υπάρχουν πολλά μέτρα που πραγματικά δημιουργούν προβλήματα και είναι μια παράδεκτη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Για το TVI, αυτό το οποίο έχω υπόψη, ποιο είναι ο συγχρονισμός του TBI. Όχι όμως ε, συνολικά, σφαιρικά και σε σχέση με τις προτάσεις που ε, θα υποβληθούν. Προσπαθούμε να δούμε αν θα υπάρξουν δυνατότητες να επιτευχθεί πρόοδος και τότε θα εξειδικευθούν οι προτάσεις μας. Αυτό και σε σχέση και με την ε, εντολή που ε, δίδεται όταν έχει γίνεται κάποιος επίτροπος ε, υπάρχει αυτή η προοπτική όμως υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι σε σχέση με αυτό το πλαίσιο η απειλή μέτρων ανταπόδοσης η, ε, μέτρων που θα επιβαρύνουν ε, η μάσα. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε μετριοπαθώς αυτά τα θέματα με τις θέσεις που υιοθετούμε. Δεν πρέπει κανείς να ε, εξαπλουστεύει τα θέματα αν είναι κανείς υπέρμαχος των ελεύθερων αγορών ή ε, υπέρ μιας προστατευτικής προσέγγισης. Ρεαλιστές πρέπει να είμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να μπορούν να λειτουργήσουν οι προτάσεις μας. Ως φιλελεύθερος λοιπόν, στρεφόμενος με πραγματιστικό τρόπο στα προβλήματα προσπαθούμε να τα επιλύσουμε με ρεαλιστικό τρόπο. Να δούμε Πώς μπορεί έτσι να επιτευχθεί πρόοδος. Άλλα θέματα για τα οποία αναφέρθηκε η παρέμβαση Κασάκα και δεν ο μόνος και ο κύριος Ντέιβιν Μάρτιν Υπάρχουν αυτά τα θέματα. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι αυτό το οποίο καταφέραμε πρόσφατα να πετύχουμε όσον αφορά το GI είναι Our partners uh, μια συμφωνία να επιτευχθεί συμφωνία και επί των GIs. Δεν μπορεί αυτό να αγνοηθεί να τεθεί στο περιθώριο και αυτό αποτελεί τμήμα των, της συμφωνίας. Όμως αληθεύει ότι οι ΙΠΑ διαφωνούν, παρότι κάνουν το ίδιο από ένα παράθυρο με, μέσω μιας άλλης δυνατότητας εμπορικά. Ναι, αλλά θεωρούμε ότι αυτά που ανέφερε ο David Μάρτιν για την πίεση αυτή σε σχέση με εταίρους που επίσης διαπραγματεύονται από αυτών των θεμάτων γιατί γίνεται η προσπάθεια από πλευρά ε, κάποιων να δοθεί μικρότερη διάσταση σε αυτό, άλλοι δίνουν μεγαλύτερη διάσταση σε αυτό. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτές τις διαφορές στη διαπραγμάτευση. Αυτό που κάνουμε είναι όμως προσπαθούμε να επιτύχουμε και σημειώνουμε σταθερή πρόοδο κύριε Καζάκα ως προς αυτά. Χωρίς να αναφερθώ σε λεπτομέρειες τώρα, πιστεύω ότι το τέλος αυτής της εντολής θα μπορέσει κανείς να κρίνει και να αξιολογήσει και να πει ότι τα GIs θα είναι αναπότρεπτα πλέον και αμετάκλητα μέρος και τμήμα αυτών των διαπραγματεύσεων. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και για τις δικές μας προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που να μπορεί κανείς ε, εις το διηναικές, στην αιωνιότητα να προστατεύει. Πρέπει να τα δούμε αυτά και σε σχέση και με τα GIs. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές λοιπόν. Αλλά μάλλον με ευχαριστεί το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Είμαι κάπως ικανοποιημένος πρέπει να πω. Επίσης ο κύριος Καζάκο επίσης ανέφερε το, το εργαλείο, το μέσο το οποίο προτείναμε όχι μόνο για το GPA αλλά και διμερός Πιστεύω ότι θα έχει επίπτωση αυτό στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο. Και για το άνοιγμα αγορών που είναι σημαντικές πρέπει να πω σε σχέση με τους εταίρους και όλας με τους οποίους διαπραγματευόμαστε. 18% περίπου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σε εταίρους στην Ασία είναι 30% ή και καμιά φορά ακόμα πολύ παραπάνω. Και δεν είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα. Έχουμε το ομοσπονδιακό επίπεδο, το κρατικό επίπεδο, περιφερειακό. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι σε σχέση με όλα αυτά η απόφαση είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι κανένας άλλος αρμόδιος για να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Τα κράτη-μέλη, συμβαλόμενα μέρη, μπορούν να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δουλειά στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να αναπτύξει νομολογικά, νομοθετικά τις προτάσεις και την περαιτέρω εξέλιξη. Δεν πρέπει προστατευτικά να υιοθετούμε κάποιες θέσεις, αλλά δεν πρέπει να είμαστε και ανόητοι και να απεμπολούμε τις θέσεις μας ελαφρά την καρδία. Αυτού του είδους οι διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις δεν διεξάγονται μεταξύ αγγέλων και αμέμπτων, αψόγων. Ένας βαθμός πραγματισμού μπορεί να είναι επωφελής καμιά φορά. Για το ηλεκτρονικό διαβατήριο, e-pass μπορεί κανείς να το φανταστεί αυτό κύριε ότι ιδιαίτερα όταν ομιλείτε με τις κρατικές αρχές με τους αρμόδιους που είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί για να μην αναφέρω κάτι περαιτέρω. Αλλά αυτό όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις μας για το ηλεκτρονικό διαβατήριο ΙΠΑΣ, αλλά στις διαβουλεύσεις με όλους. Διεξάγεται συζήτηση στο επίπεδο συνόδου κορυφής και λέγεται να υπάρξει μια συμφωνία για την Economic Partnership, εμπορική εταιρική σχέση και Economic Partnership Agreements, ε, όχι το ηλεκτρονικό διαβατήριο, αλλά Economic Partnership Agreements ε, διορθώνω. Είναι σημαντικό. Πρόκειται για το συσχετισμό μεταξύ των ε, διοικήσεων των κρατικών αρχών και των εταίρων και πρέπει να ληφθούν οι διαφορετικές θέσεις υπόψη. Αλλά υπάρχουν επίσης και ιδεολειπτικές θέσεις και θέματα ιδεολογίας που μας ε, περιορίζουν και δεν εξυπηρετούν αυτές ε, το νόημα των διαπραγματεύσεων με τις ε, εμπλεκόμενες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μπορεί όλα να εξάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά από πλευρά τους. Αλλά έχουμε και το θέμα όσον αφορά και θέματα υγείας για παράδειγμα και ασφάλειας που θα μπορούσαν να βοηθηθούν να εξάγουν πολλά περισσότερα. Επίσης πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή χρονικά θα δείτε ότι ξεκινούν αυτά τα πράγματα, μπορούν να ξεκινήσουν και να ακολουθήσουν ταχύτα τους ρυθμούς στην εξέλιξή τους. Το σημαντικό είναι να υπάρξει αυτή η απαρχή, να ξεκινήσουν, να υπάρξει αυτή η έναρξη Είμαι πρόθυμος να είμαστε ελαστικοί διότι σε ένα μακροπρόθεσμο χρονοορίζοντα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε δεν αναμένω να είναι εξίσου ελαστικές αυτές οι χώρες αυτοί οι συμβαλόμενοι όπως εμείς, αλλά πρέπει να καταλήξουν στο τι επιθυμούν, τι είναι αυτό που θέλουν πραγματικά. Δεν μπορεί να έχει κανείς και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Είναι διαπραγματεύσεις αυτές και διακυβεύονται αρκετά πράγματα. Αν θέλει κάποιος να αναπτύξει την οικονομία του, οι υπηρεσίες είναι σημαντική υπόθεση. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία χωρίς να υπάρχουν εξειδικευμένες ικανοποιητικού επίπεδου τέλειες θα έλεγα και όλας ε, δυνατότητες παροχής υπηρεσιών. Σημαντικό στοιχείο αυτό για τις οικονομίες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό και να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματικοί ως προς τις υπηρεσίες χάρη των οικονομιών τους. Για το Βιετνάμ τώρα. Στην Πνομπέν της ε, Καμπόζης συνάντησα τους ε, Βιετναμέζους εταίρους μας. Ολοκληρώσαμε το scoping exercise. Έχουμε προχωρήσει, είμαστε έτοιμοι, είναι έτοιμο αυτό τώρα. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρξει εντολή, να πάρουμε την εντολή των κρατών μελών. Ζητούμε λοιπόν να δοθεί αυτή η εντολή, εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Scoping exercise, το έγγραφο αυτό, το οποίο όσον αφορά το TPC μπορείτε και εσείς να το έχετε. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό το ότι τώρα υπάρχει αυτή η όθηση που διαμορφώνεται με τους εταίρους μας, τους Βιετναμέζους, να εμπλακούν, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και να συνεχίσουμε με επιτυχία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ε, σχετικά γοργά με αυτές τις διαπραγματεύσεις. χαιρετίζω το ότι εσείς είσαστε ο εισηγητής για αυτό το θέμα. Από πλευράς του κυρίου Ντάρτμουθ τα όσα αναφέρατε φαίνεται ότι η απάντηση στην επιστολή σας έχει προετοιμαστεί, αλλά μπορώ να σας δώσω και προφορικά την απάντηση. Δεν είναι για την, ε, τα θέματα μετανάστευσης αυτό. Είναι περισσότερο για την κυκλοφορία, ελεύθερη κυκλοφορία στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων μεταξύ πολυεθνικών ε, στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Δεν είναι θέματα μετανάστευσης ή που, κάτι που να αφορά τη μετανάστευση ξεχωριστά καθόλου. Αυτό το οποίο είχε ε, τεθεί ήταν ότι θα μπορούσε αυτό να είναι δυνατό να γίνεται από μια χώρα προς μια άλλη. Όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της επικράτειας μιας χώρας, αλλά και από μια χώρα σε μια άλλη ώστε να, ανταποκριθούν ή να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που υπάρχουν. Είναι λοιπόν θέμα υποσυζήτηση. Συζήτηση ευρύτερα και με την Ινδία τώρα. Πρόσφατα λάβαμε μια προσφορά όσον αφορά τις υπηρεσίες και είναι απογοητευτικό αυτό, είναι απογοητευτική κατάσταση. Απέστειλα μια επιστολή προς τον Ινδό ομόλογό μου λέγοντας ε, ξεκάθαρα αυτό ότι αν αυτό είναι η βάση τότε δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτό που βλέπω και χωρίς να υπησέλθω σε λεπτομέρειες είναι ότι αυτό έχει επιπτώσεις, έχει τις επιπτώσεις του όσον αφορά τις ε, κρατικές ε, ε, εκλογές, ε, περιφερειακές εκλογές, την Ούταρ Πραντές για παράδειγμα, αυτή την, αυτό, αυτό, το κρατήδιο της Ινδίας. Δεν μπορώ να επισέλθω, δεν θέλω να επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες, αλλά αυτό μπορεί να αποτελέσει τμήμα της ευρύτερης εικόνας που μπορεί να έχει κανείς. Τώρα, επιλέγοντας την καλύτερη ημερομηνία για την Market Access Regulation, θα έλεγα είναι ένα λογικό χρονοπλαίσιο. Όμως είμαι ανοιχτός να συζητήσω τα θέματα, αλλά να είναι λογικά τα πλαίσια των συζητήσεων. Δεν θα αλλάξει σε έξι μήνες ο κόσμος. Και αν αλλάξει, θα αλλάξει ανεξάρτητα από την Market Access Regulation. Αλλά με λογικό τρόπο, μέσα σε κάποια όρια και πλαίσια και μέσα σε ένα χρονοπλαίσιο ε, που θα πρέπει να μας οδηγήσει να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα για τον Καναδά. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, Πρόεδρε. Για τον Καναδά νομίζω μπορούμε φέτος να πετύχουμε μια συμφωνία. Θα έλεγα μπορεί να γίνει αυτό, ναι. Οι υπηρεσίες μας έχουν χρησιμοποιήσει, πήραν αρκετό χρόνο γιατί για πρώτη φορά ε, προσέγγισαν αυτό το θέμα με έναν κατάλογο αρνητικών θεμάτων, negative list approach, όπου θα πρέπει να υπάρξει ε, συσσόρευση όλων των θεμάτων στην κατάρτιση αυτού του καταλόγου από όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει τεράστια δουλειά, υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν, αλλά ελπίζουμε ότι πριν από τα τέλη του έτους θα κλείσει το θέμα και θα διευθετηθεί. Δεν βλέπω κάποιον λόγο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι θα αλλάξουν τόσο πολύ τα πράγματα ώστε να μην μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους. Ρωσία τώρα. Βλέποντας την συνθήκη για την προσχώρηση στον ΠΟΕ, πολλά υπάρχουν σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις και τα συναφή θέματα. Επίσης για την υγεία και την ασφάλεια επίσης. Πολλά τέτοια θέματα. η δική μου εντύπωση που έχω αποκομίσει και δεν είναι μόνο εντύπωσή μου, ελπίζω θα αλλάξουν την άποψη ότι έκαναν παραπάνω από αρκετά μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται να πάνε πιο πέρα και να κάνουν κάτι παραπάνω. Τι να κάνουμε. Σημειώνουμε, σημειώνω απλά αυτή τη θέση τους δεν αναμένεται λοιπόν μεγάλη πρόοδος τους επόμενους μήνες ή του, το επόμενο έτος όσον αφορά θέματα εμπορίου και επενδύσεων όσον αφορά τους Ρώσους. Δεν αναμένουμε κάποιες τέτοιες ριζοσπαστικές αλλαγές. Από την άλλη πλευρά τώρα, αν όλα όσα αφορούν, αφορούν αυτή την ε, συνθήκη πρόσβασης ένταξης στον ΠΟΕ εφαρμοστούν, ε, τότε αυτό δεν θα είναι ασήμαντο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ακόμα για το ETS και διάφορα άλλα τέτοια θέματα δεν είναι καθόλου εύκολο το περιβάλλον, το πλαίσιο αυτό. Αλλά η γενικότερη σκέψη τους είναι κάναμε αρκετά, πια φτάνει. Δεν το βλέπουν σαν μια ας το πω δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο πέρα. Για τις γαλλικές εκλογές δεν θα σχολιάσω το θέμα των γαλλικών εκλογών. Θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε θα είναι ο μελλοντικός πρόεδρος της Γαλλίας ως αποτέλεσμα ελεύθερων και δίκαιων εκλογών δική τους δουλειά είναι των Γάλλων να λάβουν την απόφαση ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρός τους. Ποιο κόμμα θα ψηφίσουν, ποιο πρόεδρο θα ψηφίσουν, τι θα γίνει σε σχέση με, το επόμενο, με την επόμενη κυβέρνηση. Ίσως δεν είναι κάποιοι πιο πεπισμένοι ε, υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, αλλά τέλος πάντων δική τους δουλειά είναι να αποφασίζουν ποιος θα είναι ο πρόεδρός τους. Εντάξει, λοιπόν για την άκτα τώρα. και για το θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος, πολύ σημαντικό. Μπορεί να ψηφίσει κανείς και να εγκρίνει όταν υπάρχει εκκρεμότητα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι, μπορεί να το κάνει κανείς ε, αυτό το πράγμα. Είσαστε ε, υπέρμαχος του συνταγματικού πλαισίου και έτσι πρέπει να είμαι προσεκτικός στην απάντηση που θα σας δώσω. Όμως δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το ερώτημα. Είναι περισσότερο το ερώτημα γιατί να το έκανε κανείς αυτό. Δεν υπάρχει ακόμα μια τουλάχιστον δημόσια επαρκής ικανοποιητική απάντηση. Και δεύτερον, είναι σόφρον να το κάνει κανείς αυτό. Πρώτον, γιατί θα το έκανε κανείς αυτό. Γιατί να το κάνει. Φοβάται κανείς ε, την ομολογία, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δικαστηρίου. Όχι. Θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση και για τα προβλήματα που υφίστανται εντάξει θα τα δούμε με βάση τις προτάσεις. Ευελπιστώ λοιπόν ακόμα και μετά την απόφαση όσον αφορά την, ε, ε, τον Επίτροπο για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων ακόμα και αν υπάρχουν οποιασδήποτε διαφορές πρέπει να σεβόμαστε αυτή την πτυχή. Δεύτερον, θα ήταν σόφρον κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θα ήταν. Ήμουν ένας από εσά ήμουνα επί 14 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα ε, γνωρίσει και είχαμε με τον Ντέβιν Μάρτιν δουλέψει σκληρά για να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου. Οι καλύτεροι φίλοι μας ε, στην προσπάθεια αυτή ήταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει πάμπολα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και απλά πιστεύω ότι δεν θα ήταν σόφρον λοιπόν να κάναμε κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία από πλευράς συνθήκης, πολιτικά θα έπρεπε να καταφέρουμε να την εφαρμόσουμε, ακόμα και αν θα θεωρούσαμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό όχι επειδή απεμπολεί κανείς κάποιες δυνατότητες αν υπάρχει πολιτική πλειοψηφία ακόμα και μετά από μια αρνητική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν κλείνει κάποια δυνατότητα. Θα είχε πολύ περισσότερο νόημα λοιπόν να είχαμε ένα υπόμνημα, μια γνωμοδότηση, μια έκθεση αποσαφηνίζοντας τις απόψεις μας επ' προβληματίστηκα και όχι μόνο προβληματίστηκα αλλά και συζήτησα και με εκπροσώπους των υπηρεσιών μας, των γενικών μας διευθύνσεων. Υπάρχει κάποιο πραγματικό πρόβλημα με την άκτα. Ναι, πολιτικά υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα προφανώς. Όντως, πολύ περισσότερο για τις ευαισθησίες ε, κάποιων πλευρών. Αλλά αυτό συμβαίνει και με, τις, με τα περισσότερα προβλήματα. Μπορεί να επιληθεί. Πιστεύω μπορούν να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, για το σύνολο των θεμάτων που τίθενται υπό συζήτηση, δεν θα τα επαναλάβω όλα αυτά, για την εμπορική κλίμακα και των θεμάτων αυτών και τις επιπτώσεις. Είναι σαφής ε, ε, η κατάσταση. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να διαβάζουν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Ευρωπαϊκή Κλίμακα και τις επιπτώσεις. Πολύ περισσότερο λοιπόν πρέπει να έχουμε σαφείς απόψεις για το πού θέλουμε να κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να επανέλθουμε με απαντήσεις. Δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω και σημαίνει και αυτή ότι το πολιτικό περιβάλλον απλά δεν προσφέρεται για να έχουμε μια τελική ψήφιση επ' αυτού, όντας ε, ε, ένα ε, θεμελιώδες θέμα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ίσως όμως εδώ και κάποια κενά, παράθυρα. Δεν είναι θέμα υπογραφής εν λευκό ε, μιας επιταγής ε, και μετά να δούμε το θέμα του ε, ουσιώδους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συνάδελφοί μου πρέπει να δουν τις προτάσεις σε σχέση με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, να δούμε τις πτυχές όσον αφορά την ε, επιβολή των ε, διατάξεων για το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά θα είναι ε, τα σημαντικά, η σημαντική ακρογωνιαίοι σημαντικη ακρογωνιαί λυθη για μια ουσιαστική πρόταση που θα υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους ή του χρόνου για να μένουμε επίσης και την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού αυτό. Και στο μεσοδιάστημα έχουμε ημίχρονο μου φαίνεται ότι αυτή είναι η πιο λογική πρόταση. Όμως το Ευρωκοινοβούλιο εν τη σοφία του, αν έχει άλλη άποψη, το σεβόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά όμως ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση που θα έπρεπε να υιοθετηθεί όσον αφορά την πιο σοφή προσέγγιση για την επίλυση του θέματος. Σας ευχαριστούμε, uh, Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή δημόσια συνεδρίαση. Έχουμε όμως και μια συνεδρίαση κυκλισμένων των θυρών με τον Επίτροπο. Όποιοι λοιπόν... Α, δεν μου επιτρέπετε, λέει ο κύριος Τεχούχτη, η κυρία Ρόφολ, είχε κάνει κι άλλο ένα ερώτημα για τη στάση των ΗΠΑ. Δεν έχω καταθέσει ακόμα το πώς το λένε. Α, τα μέσα επικύρωσης, instruments of ratification. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει. Αν θα το κάνω χωρίς εμάς δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει νόημα, γιατί αν δεν είσαι σε μια συμφωνία δεν έχει νόημα. Ο πρόεδρος, λοιπόν, εδώ, παραλαμβάνω, ολοκληρώνει τη δημόσια συνεδρίαση. Παρακαλώ όσοι δεν έχουν εργασία να αποχωρήσουν. Please.